Καλησπέρα σας. Ε, περιμέναμε για 10 λεπτά για λόγους ευγένειας, περισσότερο δηλαδή από ό,τι κανονικά θα έπρεπε. Οπότε ας ξεκινήσουμε άμεσα τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καταρχήν έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και σε σχέση με την πρώτη εκδοχή που λάβατε. Υπάρχει μια πρόταση τροποποίησης σε σχέση με την ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Ρωμέβα για το πολιετές ε, σχέδιο, ε, σχέδιο ανάκτησης του τόνου του Ατλαντικού και άρα θα το αναβάλουμε για την συνεδρίαση της 22ης Ιανουαρίου. Έχετε κάποια ερώτηση? Αν όχι, θα το κάνουμε αυτό και έτσι αλλάζουμε την ημερήσια διάταξη και αφαιρούμε αυτήν την ψηφοφορία. Στις ανακοινώσεις του Προέδρου έχω να σας πω, να σας ξαναπώ, ότι όταν τελειώσει η απόψινή συνεδρίαση θα μετακομίσουμε Δηλαδή θα πάμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και το καινούριο χρόνο θα έχουμε την ευκαιρία να πιούμε όλοι παρέα ένα ποτηράκι στις 6.30 στο 5 Ζ. Και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι εκεί. Και περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η δημόσια κρόση για την αξιολόγηση της ε, ε, του αλευτικού κανονισμού για τη Μεσόγειο. Έχουν περάσει 7 χρόνια από την έναρξη ισχύου του κανονισμού αυτού που ισχύει και εφαρμόζεται για την αλία στη Μεσόγειο. Έχετε όλα τα έγγραφα και τις μελέτες που έχουν γίνει για αυτό το θέμα και ε, υπάρχουν και στην εφαρμογή e-meeting. Έχουμε οργανώσει αυτή την ακρόαση σε δύο χωριστά κομμάτια, δύο χωριστά τμήματα. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην περιγραφή της κατάστασης των λευτικών πόρων στη Μεσόγειο και στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Και το δεύτερο τμήμα αφορά αυτή καθ' αυτή την αξιολόγηση του κανονισμού περιαλίας στη Μεσόγειο. Έχουμε εμπειρογνώμονες από το κοινό κέντρο έρευνας και στο δεύτερο τμήμα θα ακούσουμε την Κομισιόν αλλά και μια μη κυβερνητική οργάνωση καθώς και εκπροσώπους του αλευτικού τομέα. Σας χαιρετίζω ήδη όλους και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα παρόντες εδώ και για τη συνεργασία σας για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Και αν θέλετε, επειδή ήδη έχουμε αρχίσει λίγο, χωρίς άλλα προήμια, να ξεκινήσουμε με το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας. Καλώ τον κύριο Τζάκομο Όσιο από το Κοινό Κέντρο Έρευνας να μας παρουσιάσει την κατάσταση των βασικών ελευτικών πόρων στην Μεσόγειο. Και όπως πάντοτε, από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί η παρέμβασή σας, θα έχουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων Κύριε Όσιο, έχετε λοιπόν τον λόγο. Καλώς ορίσατε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω μια επισκόπηση της κατάστασης ε, των αληθικών παρών στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Εκείνη προσπάθεια με τον Μαξιμιλιάνο Καρδινάλη, ο οποίος εργάζεται στο Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γερικών Επιστημών. Η δουλειά μου είναι στο Κοινό Κέντρο Ερεύνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάποιοι συναδελφοί μου ήταν εδώ πριν από δύο εβδομάδε και παρουσίασαν το θέμα των ενισχύσεων στον τομέα της αλληλείας ε, και συζήτησαμε το θέμα της ε, απόδοσης των επενδύσεων. Λίγα πράγματα από επιστημονικής απόψεως και μετά τα αποτελέσματα της αξιολόγηση των αποθεμάτων. Θα προσπαθήσουμε τέλος να ερμηνεύσουμε τις τάσεις, την ελληνική προσπάθεια και εν συνεχεία θα γίνει ανάλυση κινδύνου των εκτιμωμένων αποθεμάτων και θα καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας. Από πλευράς ορολογίας θα συζητήσουμε σήμερα τον όρο SSB, δηλαδή την βιομάζα των ενηλίκων ψαριών σε αναπαραγωγική ηλικία. Επίσης τη θνησιμότητα, το F είναι η θνησιμότητα λόγω αλίευσης και το FMSY, Maximum Sustainable Yield, είναι το F, λαμβανωμένης υπόψη της μακροπρόθεσμης απόδοσης και της μεγιστοποίησης της αηφορικής εκμετάλλευσης των αποθεμάτων. Σήμερα θα εξετάσουμε κυρίως τον λόγο μεταξύ του F για την τελευταία χρονιά εκτίμησης και, το FMS, και του FMSY. Ο λόγος αυτός ακριβώς μας δίνει και το πόσο μακριά είμαστε από τον επιθυμητό στόχο, το FMSY. Εάν ο λόγος αυτός είναι μεγαλύτερος από ένα, σημαίνει ότι το απόθεμα υφίσταται εκμετάλλευση. Το αντίθετο συμβαίνει για την τιμή κατά από ένα. Η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα υποδιαιρούνται σε 30 υποενότητες από στρατιστικής απόψεως βάσει ακριβώς των ορισμών της ε, Επιτροπής Ελίας για τη Μεσόγειο. Οι περισσότερες εκτιμήσεις γίνονται με βάση αυτήν την υποδιέρεση της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Σήμερα θα σας δώσω και θα συζητήσουμε κυρίως τις εκτιμήσεις που αφορούν τα ευρωπαϊκά είδετα δεδομένου ότι δεν γίνονται και πολλές εκτιμήσεις για την Νότιο Μεσόγειο. Εν γέννη, η Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή, η ΣΤΕΚΦ από το 2008, μελετάω και περισσότερα είδη. Δεν έχουμε σημεία αναφοράς για τα περισσότερα ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε καλές προσεγγίσεις. Αυτή τη στιγμή μελετούμε 40 με 50 αποθέματα τον χρόνο. Δύο λόγια για την διαδικασία, για να καταλήξουμε σε κάποια εκτίμηση αποθέματος. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα που βγήκαν από λίγο πολύ πέντε έτη εκτιμήσεων. 16 εμπειρογνώμονες της ΣΤΕΚΦ e δουλεύουν πάνω στο θέμα. Όλες αυτές οι εκτιμήσεις αξιολογήθηκαν από την ΣΤΕΚΦ. E Στοιχεία της DCR πήραμε επίσης μέχρι το 2008 και από την DCF αυτά τα δεύτερα για την περίοδο 2002-2012. Αυτά τα συνέλεξε το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την συλλογή των δεδομένων κατά τη διάρκεια 12 περίοδων συλλογής. Η εκτίμηση γίνεται κάθε χρόνο ουσιαστικά κάθε απόθεμα και αυτά εξετάζονται από την αντίστοιχη ομάδα εργασία τη Επιτροπή Ελία για τη Μεσόγειο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο όγκο ποιοτικών αξιόπιστων σταριστικών δεδομένων που είχαμε ποτέ στη διάθεσή μα για την Μεσόγειο. Αν πάμε στα πρώτα αποτελέσματα, βλέπετε εδώ ένα διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η εκμετάλλευση μια συγκεκριμένη χρονιά και συγκρίνεται με τον λόγο F, FMSY. Τα παθέματα πάνω από τη γραμμή, τη χάνουν υπερεκμετάλλευσης. Αυτά που είναι κάτω είναι σε υφορική κατάσταση. Θεωρητικά, εάν η γραμμή αυτή την οριζοντιωθεί σημαίνει ότι έχουμε πιο αεφορική διαχείριση. Αν τα δούμε αυτά έτος προς έτος, από το 7 ας πούμε στο 2012, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κλίση και αυτό πιθανότητα σημαίνει ότι εν γέννη δεν σημειώνεται βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων. Αν δούμε τώρα κάποια αποτελέσματα με μεγαλύτερη ανάλυση, ειδού τα αποτελέσματα της περαιτέρω ανάλυσης της ΣΤΕΚΦ μεταξύ 2008 και 2012. Κάθε επιτροπή εδώ εκπροσωπεί τις διάφορες στατιστικές ομάδες Βλέπετε εδώ τις βαλερίδες τον κόλπο της ε, Λιών, την, τον Τυρινικό κόλπο, το 11 είναι η Σαρδινία. Βλέπετε λοιπόν διάφορες περιοχές εδώ. Ε, η Νότια Σικελία, η Μάλτα. Εν γέννη. Και πάλι η ίδια εικόνα. Σχεδόν όλα τα αποθέματα και τα αποθέματα για τα οποία έχουμε εκτίμηση τη χάνουν υπερ-εκμετάλλευσης. Βλέπετε μάλιστα την απόσταση από το 0. Το 0 είναι το FMSY, η εφορική, το εφορικό απόθεμα. Σε άλλες περιοχές είναι η 16 έως 29 Νέα Νότια Ιταλία, Αδριατική, 17 συγκεκριμένα, το 18 είναι η Νότιος Αδριατική, το 19 είναι η Νότιος Ιταλία, το 20, 22 και 23 ε, είναι τα ελληνικά κατά κύριο λόγο είδετα. Στην Ελλάδα θα παρατηρήσετε ότι δεν έγινε εκτίμηση μετά το 2008. Δεν συλλέξαν δηλαδή στοιχεία μετά το 2008. Και τέλος, το 25 είναι η Κύπρος και 29 είναι η Μαύρη Θάλασσα, ο εύξηνος πόντος. Όπως βλέπετε, υπερεγμετάλλευση των περισσότερων αποθεμάτων με κάποιες εξαιρέσεις. Αυτά θα το ομαδοποιήσουμε εν συνεχεία σε κάποια διαφάνεια για να δείτε πώς ε, αποτυπώνονται όλα μαζί. Η Σαρδέλα βλέπουμε εδώ ότι στην περιοχή 16 τη χάνει εφορικής εκμετάλλευσης, ο Γάβρος στην 17, κάποια άλλα αποθέματα τη χάνουν εφορικής ε, εκμετάλλευση στην Ελλάδα, στην περιοχή 20 και κάποια μπαρμπούνια το ίδιο. Αν δούμε τώρα τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αποθεμάτων από την Επιτροπή της Μεσογείου βλέπουμε ότι έχουν καταλήξει λίγο πολύ στα ίδια αποτελέσματα. Συγκλίνουν λοιπόν οι εκτιμήσεις από τα δύο όργανα Αν βασιστούμε πάντως στις εκτιμήσεις της ΣΤΕΚΦ και ονοματοποιήσουμε τα αποθέματα ανά ομάδες ειδών θα δούμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σαφή στάση ως προς το ποια είδη δηλαδή τι κάνουν υπερεκμετάλλευση και πια όχι. Ας πούμε στα βαθύβια. Σχεδόν όλα τα αποθέματα τη χάνουν υπερεκμετάλλευση. Με πέντε μόνο εξαιρέσεις. Όσον αφορά τα οστρακόδερμα, το Παρπενέους Λαγκινόστρις και το Νέφροψ είναι τα μόνα τα οποία εκτιμήθηκε ότι την χάνουν αεφορικής εκμετάλλευσης. Όλα τα άλλα και πάλι αλλιεύονται. Τα μοναμαλάκια με το οποία ασχοληθήκαμε ήταν το χταπόδι και αυτό την χάνει υπερεκμετάλλευσης. Είναι μικρά παλαιγικά είδη. Η κατάσταση είναι μάλλον ανάμεικτη. Τα τρία αποθέματα που λέξαμε είναι η Γαβροσαρδέλα, και ένα είδο. Εκεί η εικόνα είναι ανάμεικτη, όπω είπα. Είναι μισά-μισά περίπου. Τα ίδια όσον αφορά την υπερεκμεταλλευσή του, την υπεραλίευσή του. Αυτέ είναι εκτιμήσει όσον αφορά τα αποθέματα. Όλα αυτά ε, τα έχουμε αξιολογήσει. Είναι αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό είναι κομμάτι τη δικής μου δουλειά με τον Μαξ Καρδινάλε. Τι κάναμε εδώ. Καταγράψαμε τις τάσεις στην αληφτική προσπάθεια. εστιάζοντας α, κυρίως τις σειρόμενες στράτες βυθού με παράθυρο με πόρτες ε, μετρήσαμε τις α, ημέρες επί κιλοβάτ συγκεκριμένα και εδώ βλέπετε ποια είναι η συμβολή της ελληνικής προσπάθειας της κάθε χώρας στο σύνολο. Και βλέπετε τις επιμέρους τάσεις, αναχώρα δηλαδή. Η Ιταλία σε αληθική προσπάθεια είναι πρώτη, η Ελλάδα είναι αρκετά ψηλά θα λέω. Μετά έχουμε την Ισπανία και Γαλλία, Μάλτα, Κύπρος, Σλοβενία πιο κάτω. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στην Ιταλία αλλά και στη Γαλλία. Βλέπετε σημαντική πτώση. Αυτά είναι στοιχεία του 2012. Εάν πάμε σε λίγο μεγαλύτερο βάθος για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει ακριβώς σε κάθε περιοχή συλλογής στατιστικών δεδομένων, βλέπουμε ότι στην Ιταλία στην περιοχή 10, 11, 16, 17 και 18 βλέπουμε ότι εκεί η προσπάθεια πέφτει. Α, και στην περιοχή 9, ενώ στη 19 έχουμε μια μικρή αύξηση, ένταση. Αυτά για την περίοδο 2004-2012. Στην Ισπανία η τάση είναι πτωτική εν γέννη. Όμως, αν ρίξουμε και πάλι μια καλύτερη ματιά στα ίδια στοιχεία, για να δούμε αν υπάρχει εφοροποίηση μεταξύ επιμέρους στόλων. Εδώ βλέπετε τα πρωτογενή δεδομένα. Ανά περιοχή συλλογή στοιχείων. Βλέπετε εδώ το μήκος του σκάφους με ροζ ε, είναι τα μεγαλύτερα, μεγαλύτερες στράτες. Βλέπουμε λοιπόν το μέγεθος αυτό εν γέννη τίνει να μειωθεί. Φαίνεται ότι σε προσπάθεια και οι μικρομεσαίες στράτες πέφτουν σε προσπάθεια. Εδώ μας βλέπετε στην περιοχή 6 και στην 5 ήταν οι Ισπανικές τράτες στον ε, κόλπο του Λέοντα και εκεί έχουμε μια ένταση της προσπάθειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει περισσότερο, περισσότερη διερεύνηση. Δεν ξέρουν πού οφείλεται. Γιατί μπορεί η ένταση, η ελιστική προσπάθεια αυτού του τμήματος του στόλου να έχει ενταθεί και τα νούμερα να μην αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματικότητα. Στην Ιταλία κάνουμε τους ίδιους υπολογισμούς και φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα σκάφη μειώνονται σε πλήθος ενώ τα μεσαία σε μέγεθος σκάφη παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση σε κάποιες περιοχές ή παραμένουν σταθερά. Κάπου αλλού έχουμε και μερικές μικρές μειώσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι η προσπάθεια μείωσης της ελληνικής ικανότητας είναι ικανοποιητική για να πετύχουμε το περίφημο FMSY. Πετυχαίνουμε λοιπόν εφορική εκμετάλλευση ή όχι. Εδώ βλέπετε παλαιότερα αποτελέσματα εκτίμηση αποθεμάτων και βλέπετε πόσο η θνησιμότητα θα έπρεπε να μειωθεί για να πετύχουμε την FMSY. Εδώ για όλα τα εκτιμωμένα αποθέματα. Ας πούμε για τον Μερλούκιο στην περιοχή 7 η ελευθερική προσπάθεια θα έπρεπε να μειωθεί κατά 86% για να πάμε σε εφορική κατάσταση. Βλέπετε λοιπόν ότι απαιτούνται πολύ ψηλά ποσοστά μείωσης για τα περισσότερα αποθέματα. Στην περίπτωση της ε, γαρίδας που πάει καλά στην περιοχή 9 βλέπετε ότι θα μπορούσε κανείς να αυξήσει και την ελευτική προσπάθεια γιατί είμαστε μακριά από το FMSY, την εφορική ελευτική προσπάθεια. Το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές Βλέπετε εδώ ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να μειωθεί το F, πρέπει να μειωθεί η ελευθερική προσπάθεια. Όλα αυτά βεβαίως βάσει των στοιχείων της ΣΤΕΚΦ. που λίγο πολύ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο 85% των περιπτώσεων μέχρι και το 12% η εκμετάλλευση αυτών των αποτυμάτων δεν ήταν εφορική, δεν ήταν βιώσιμη. Έχουμε εδώ και άλλα αποτελέσματα της ΣΤΕΚ. Βλέπουμε ότι απαιτείται και εδώ μεγάλη σημαντική μείωση. Έχουμε και μερικά πελαγικά είδη εδώ, λίγα όμω, αλλά με πάση περιπτώσει η κατάσταση και πάλι η εικόνα δεν αλλάζει. Το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, είναι το ίδιο, ότι 90-95% των αποθεμάτων που αναλύσαμε φαίνεται ότι την χάνουν μεταξύ 2010 και 2012 μη αεφορικής, μη βιώσιμη εκμετάλλευσης. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες εργασίας της ΤΕΚΦ, προέβησαν σε μοντελοποίηση κάποιων στοιχείων. Στην περίπτωση της γλώσσας, για παράδειγμα, έγινε εκτίμηση του αποθέματος στην Αδριατική. Εκεί χρησιμοποιήσαμε κάποιες νέες μεθόδους μοντελοποίησης όπου μπορεί να εκτιμηθεί η θνησιμότητα με βάση τα προφίλ διαφορετικών στόλων. Επίσης έχουμε τις ε, εκφορτώσεις από το παρελθόν που λάβαμε επίσης υπόψη μας και τα καταχωρήσαμε, τα σωματώσουμε στο μοντέλο Έτσι νομίζω ότι προσεγγίσαμε περισσότερο την πραγματικότητα. Κάναμε τα στοιχεία μας πιο αξιόπιστα. Άρα, κλείσαμε με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, ειδού τα αποτελέσματα 80 εκτιμήσεων αποθεμάτων, 24 ήδη κάλυψε η ΣΤΕΚΦ και 25 το Συμβουλίο για τη Μεσόγειο η Επιτροπή μάλλον για τη Μεσόγειο. 80 είδη, στην μία περίπτωση αφορούν ουσιαστικά ένα ζεύγος είδους περιοχής. Αυτό είναι μία εκτίμηση. Πάντως ε, στην πραγματικότητα τα, τα είδη από μόνο τους τα οποία καλύψαμε δεν είναι πάνω από 25. Αλλιώς είχαμε επαναλαμβάνω συνδυασμούς είδους περιοχής. Στη Μεσόγειο υπάρχουν 100 διαφορετικά αποθέματα που αξιοποιούμε. Καλύψαμε λοιπόν ένα μικρό αριθμό αποθεμάτων. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα άλλα αποθέματα που δεν εκτιμήσαμε στο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Το βέβαιο είναι ότι βάσει της κοινή αλληλευτικής πολιτικής τα αποθέματα αυτά πρέπει να τύχουν βιώσιμης αλήψης. Στο Κοινό Κέντρο Ερευνών προέβημε σε ανάλυση κινδύνου για να μετρήσουμε τον δυνάμει κίνδυνο για τα αποθέματα τα οποία δεν εκτιμήσαμε. Πρόκειται για μια ημι ποσοτική μέθοδο η οποία αξιοποιεί μια μέθοδο βαθμολογίας που αποτυπώνει τα εξή. Το ένα είναι η παραγωγικότητα, δηλαδή πόσο παραγωγικό μπορεί να είναι ένα αλίευμα, ένα απόθεμα και το άλλο είναι ένας παράγοντας ευαισθησίας, ευπάθειας, ο οποίος μας λέει σε ποιο βαθμό ένα απόθεμα είναι ευάλωτο, ευπαθές. βάσει του κύκλου, ε, του κύκλου ζωής, του παρελθόντων στοιχείων. Το τελικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε δηλαδή, είναι να καταλάβουμε πού βρίσκονται τα εκτιμηθέντα είδη στο συγκεκριμένο διάγραμμα. Μετά έχουμε είδη τα οποία έχουν υψηλή ευπάθεια και χαμηλή παραγωγικότητα. Αυτά είναι στην κόκκινη περιοχή. Είναι η περιοχή υψηλού κινδύνου. Ένα βέβαια στο μπλε σκούρο είναι η χαμηλή ευπάθεια και η υψηλή παραγωγικότητα. Εφαρμόσαμε τη μέθοδο αυτή σε 150 είδη πελαγικά και βενθικά συγκρίνοντας τις δύο αυτές παραμέτρους. Βλέπουμε λοιπόν τις ε, κουκίδες αυτές που είναι σωμερός σχετικά κατανεμμένες. Με τον τρόπο αυτόν βλέπουμε ποια είδη είναι στον χαμηλό κίνδυνο, δεν έχει πολλά. Στον μέσο κίνδυνο έχουμε αρκετά ζευγή είδους περιοχής και στον ψηλό κίνδυνο έχουμε βέβαια αυτά τα οποία κίνδυναν περισσότερο. Στο πλαίσιο της ανάλυσης συμπεριλάβαμε τα είδη τα οποία εκτιμήσαμε βάσει ανάλυσης προσθέτοντας δίπλα και τον λόγο F προς FMSY. Αυτό αντικατοπτρίζει τον ε, όλο ένα κίνδυνο. Μας λέει με άλλα λόγια το διάγραμμα ότι τα είδη με τους υψηλότερους ε, ρυθμούς ε, κινδυνεύουν περισσότερο και το αντίστροφο προς την άλλη κατεύθυνση. Η πληροφορία, το μήνυμα αν θέλετε που βγαίνει από αυτό το διάγραμμα είναι το εξή. Ότι όταν τα αποθέματα εκτιμώνται ποσοτικά και μετρηθούν ως μεσαίου κινδύνου, όταν είναι κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, Τότε τα αποθέματα προς τα δεξιά μπορεί στην πραγματικότητα να υπόκεινται σε ακόμα χειρότερες συνθήκες εκμετάλλευσης, να κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Αυτή είναι η, η κατάρρεξη πάντως με βάση τον κίνδυνο. Θα δούμε πού πηγαίνουν τα μεν και τα δε. Όλα αυτά ούτως ή άλλως ως μελέτη είναι στο αρχικό τους στάδιο. Πάνω στα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουμε το επίπεδο εκμετάλλευσης, εξυπηρέτηση αυτών των ελιευμάτων και να δούμε πώς θα πάρουμε μέτρα κατά της υπεραλίευσης. Με βάση την GSUN ε, ταξινόμηση αν συγκρίνουμε παραγωγικότητα και ευπάθεια Βλέπουμε εδώ πια είδη είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Βλέπετε ότι ο υψηλός κίνδυνος συνήθως πηγαίνει με την υψηλότερη ευπάθεια κατά Αγίος Ιάννη. Βλέπουμε επίσης εδώ ότι τα παθήματα που κινδυνεύουν περισσότερο είναι έλας με τον βράχια και αυτό δεν είναι έκπληξη διότι αρκετές μελέτες δείχνουν ότι στην Αδριατική έχουμε 94% μείωση σε σχέση με την δεκαετία του 40 και έλας με τον βράχια. Είναι λοιπόν είδη τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Εν κατακλείδη, μετά από τα διαγράμματα τα οποία είδαμε, θα έλεγα ότι η τελευταία, στα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πρώτον η κατάσταση όσον αφορά τις γνώσεις που χρειαζόμαστε για τα αποθέματα στην περιοχή μας βελτιώνεται γρήγορα, ταχύτατα, καλό είναι αυτό. Διαπιστώσαμε όμως ότι 94-95% των αποθεμάτων που αναλύσαμε τη χάνουν υπερεκμετάλλευση σε σχέση με το FMSY και για να επιτευχθεί, το οποίο για να επιτευχθεί πρέπει η μειώση στην αλληλευτική προσπάθεια να είναι μεταξύ 45% και 51% που έλειφθηκε η προσπάθεια. Φυσικά αυτό διαφέρει από πόθημα σε απόθεμα, γιατί μιλάμε για μεγάλες μειώσεις. Τώρα, με βάση αυτά τα οποία είδαμε όσον αφορά την ανάγκη μείωσης της ελευθερικής προσπάθειας, βλέπουμε ότι κάτι έγινε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Η ονομαστική προσπάθεια, ξέρετε, δεν είναι η καλύτερη αποτύπωση των τάσεων όσον αφορά τη θνησιμότητα των ψαριών, των αλλιευμάτων εν γέννη. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν μειώσαμε επαρκώ την ελληνική προσπάθεια ώστε να έχουμε αποτέλεσμα και στην θνησιμότητα. Αυτό θα το μελετήσουμε και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε πώ συσχετίζεται το F με την αλληλευτική προσπάθεια. Μια άλλη σημαντική πτυχή του θέματος και πάλι αυτό προκύπτει από μελέτη των Νικολικό και του 7. Φαίνεται ότι ακόμη και αν μειώσουμε την ελληνική προσπάθεια, το F, δεν θα φτάσουμε την αηφορική, το αηφορικό επίπεδο χωρίς να βελτιώσουμε και την επιλεξιμότητα, την μάλλον εκλεκτικότητα. Τι εννοώ. Σήμερα τα περισσότερα αποθέματα συμπεριλαμβάνουν, συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες ηλικίες ομάδες ψαριών. α πούμε, πολύ νεαρά άτομα, τα οποία δεν προλαβαίνουν ακριβώ να αναπαραχθούν. Οπότε, στη σχετική προσωμείωση, βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε μέσω της ρύθμισης των δικτυών να έχουμε μεγαλύτερα ψάρια στο νερό. Έτσι εισάγουμε μια νέα τιμή του F, μια τιμή αναφοράς. που λαμβάνει υπόψη της το μέγεθος του ψαριού. Και καταλήγουμε σε έναν επανυπολογισμό του μέγεθους του ψαριού με βάση μια πιο εκλεκτική μέθοδο. Είναι η στικτή γραμμή. Η συνεχής γραμμή είναι το FMSY Και μετά βλέπουμε και την απόδοση η οποία θα προέκυπτε εάν τα αποθέματα υπέκυντο σε ιδανική αλίευση. Έτσι και η απόδοση τελικά θα είναι υψηλότερη από σήμερα. Η οικονομική απόδοση επίση θα είναι πολύ υψηλότερη γιατί θα ψαρεύουμε και μεγαλύτερα ψάρια, τα μεγαλύτερα ψάρια πολλούνται σε υψηλότερε τιμέ στι περισσότερε αγορέ. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα για τα διάφορα αποθέματα. Ας πούμε λοιπόν ότι οι άμεσε δράσεις που απαιτούνται για να πετύχουμε το FMSY, την εφορική εκμετάλλευση, είναι να μειώσουμε το F για όλα τα βαρυθικά είδη, την πραγματική προσπάθεια αυτό είναι το βασικό μήνυμα προκειμένου. Επίσης, για τα πελαγικά να εφαρμοστεί ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα, ένα τάκ. Εδώ γίνεται μια πρόοδος. Είχε ξεκινήσει με τα μικρά πελαγικά. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης των συγκεκριμένων ειδών και επίσης την επιλεκτικότητα των ε, αληθικών εργαλείων. Ε, αυτό, η προσαρμογή των αληθικών εργαλείων θα μας επέτρεπε να πάμε πιο κοντά, να έρθουμε κοντά στο MSY. Μετά έχουμε και κοινέ αληθικές προσπάθειες με τρίτες χώρες. Θα χρειαστεί και εκεί να προβούμε σε εκτιμήσεις ε, αποθεμάτων. Οπότε δρόμος από εδώ και πέρα αυτό υποστηρίζουμε με βάση αυτές τις εκτιμήσεις είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε και ολοκληρωμένε εκτιμήσεις θεμάτων για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Ο αριθμός των ειδών που εκτιμούμε Πρέπει να αυξηθεί, πρέπει να κάνουμε περισσότερες εκτιμήσεις, ποσοτικές εκτιμήσεις και ιδιαίτερα για τα είδη για τα οποία λείπουν στοιχεία. Το θέμα να κάνουμε ανάλυση όπως κάναμε το PSA και από εκεί πέρα να αξιοποιήσουμε και μια ομάδα του ΦΑΟ και τη δουλειά τη, η οποία έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά και την βιομάζα αυτή καθ' αυτή, την υφιστάμενη και την ε, βιομάζα αναφοράς, η οποία επιτρέπει αεφορική διαχείριση. Τι άλλο τώρα. Από τις τελευταίες εκτιμήσεις φαίνεται ότι υπάρχουν μηνύματα ότι τα προβλήματα μειώνονται κατά κάποιο τρόπο αν και έχουμε μεγάλα προβλήματα συλλογή στατιστικών δεδομένων στην 11, στη Σαρδινία για παράδειγμα εκεί φαίνεται ότι η δημοτοληψία δεν έγινε σωστά στην Κορσική επίσης, στην GSA 8 εκεί δεν έχουμε καθόλου στοιχεία και αυτό μας ανησυχεί βεβαίω. στη Μαύρη Θάλασσα να έχει ικανοποιητικά η δειγματοληψία σε διάφορες χώρες. Για το μέλλον θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του DCF. Πέρσι το καλοκαίρι ε, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία δεν έγιναν ε, έρευνες ας πούμε, για πελαγικά είδη μεταξύ άλλων. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει και στην Ιταλία το 2013 για τις εκφορτώσεις. Σίγουρα έχει μειωθεί έτσι η δυνατότητά μας με βάση όλα αυτά να αξιολογούμε, να εκτιμούμε τα αποθέματα. Οπότε για να κλείσω, να πω ότι η παρουσίαση αυτή δεν θα έχει γίνει δυνατή αν δεν μας είχαν στείλει τα στοιχεία του στα κατημέλη. Ε, το ίδιο ισχύει για την ομάδα διαχείρισης του Κοινού Κέντρου Ερευνών χωρίς την ΣΤΕΚ βεβαίω και χωρίς τις ε, εκτιμήσεις, όπως είπα, του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Ευχαριστώ πολύ. Muy bien, muchas gracias al señor Ocio. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Όσιο για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εισήγηση και όπως συνηθίζουμε θα αρχίσουμε τώρα με έναν γύρο παρεμβάσεων ε, ερωταπαντήσεων των βουλευτών που το επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Μάλιστα, Κύριο Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Μια πολύ σύντομη και συγκεκριμένη ερώτηση. υπάρχουν κάποια αποθέματα που καλύπτονται από προγράμματα διαχείρισης. Δεν έχει υπάρξει αποκατάσταση με βάση τις πρωτοβουλίες στον τομέα αυτών. Δεν νομίζω ότι εξετάστηκε αυτό συγκεκριμένα. Εγώ θα απαντούσα ότι ίσως τα σχέδια διαχείρισης δεν έχουν εφαρμοστεί για αρκετό χρονικό διάστημα για να δούμε αποκατάσταση. αλλά ίσως αυτό να εξεταστεί τα προσεχή χρόνια. Η κυρία Λοβέν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Είναι ανησυχητική η κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αποθέματα για τα οποία δεν έχει γίνει αξιολόγηση, ενώ το 95% αυτών ε, για τα οποία έχει γίνει αξιολόγηση αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μείωση της θνησιμότητας στα αποθέματα αυτά κατά 50% περίπου. Όσον αφορά τα αποθέματα όπου δεν έχει γίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζουμε. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι προσέγγιση θα προτείνατε για τα αποθέματα αυτά μέχρι να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο τα αποθέματα αυτά τη στιγμή που δεν έχουμε αρκετά δεδομένα. Και μπορεί να μου διέφυγε, αλλά ίσως μπορείτε να μας πείτε πόσα θέματα δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα. Και βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη νέα προσέγγιση. Μιλάτε όχι μόνο για μείωση αλλιευτικής προσπάθειας, αλλά και τροποποίηση της επιλεξιμότητας για να επιτευθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρό τρόπο. Έχουμε ανάλογους υπολογισμούς στη Βαλτική για τον Γάδο. Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί. Ευχαριστώ η κυρία Φράγα. Και μετά θα δώσω το λόγο πάλι στον ομιλητή να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλώ κυρία Φράγα. Ε, ε, Είδαμε μείωση της ε, θνησιμότητας από το 55 στο 55 στο 51% στο MSY για να φτάσουμε στο MSY. Αλλά πότε, πότε θα το επιτύχουμε. Δεν έχετε βάλει πότε για το 2015 μιλάτε, 2020. Ποια ημερομηνία προβλέπετε να υπάρξει αυτή η μείωση του 45 με 51%. Ευχαριστούμε κυρία Φράχα. Άλλη παρέμβαση. Να δώσουμε το λόγο αν όχι στον κύριο για να απαντήσει. Thank Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω ανάποδα, από την τελευταία. Ο αριθμός των αποθεμάτων που δεν έχουν αξιολογηθεί δεν έχω ακριβή αριθμό και βέβαια εξαρτάται από την ε, σημασία όσον αφορά τις εκφορτώσεις του κάθε αποθέματος. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για 70-80 αποθέματα. Αλλά είναι ε, χοντρός ο υπολογισμός αυτός. Ε, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή αριθμό. Τι να κάνουμε τα αποθέματα αυτά. Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ επιστήμονας είμαι, δεν μπορώ να σας πω για τη διαχείρισή τους, αλλά Σίγουρα θα πρέπει να αναλυφθεί δράση ώστε να γίνει κάτι τουλάχιστον για τα πιο ευάλωτα αποθέματα. Υπάρχουν περιοχές με πολλαπλά αποθέματα και όπου υπάρχει η τάση η μέγιστη βιώσιμη απόδοση να υπολογίζεται σύμφωνα με το πιο ευάλωτο απόθεμα, κάτι το οποίο μειώνει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και για πιο παραγωγικά αποθέματα, αλλά βέβαια αυτό είναι κίνητρο για τους αλληλείς να βελτιώσουν την επιλεξιμότητα και να αποφύγουν τις περιοχές όπου υπάρχουν πιο πολλά ευάλωτα είδη. Ίσως όμως, και αυτή είναι προσωπική μου γνώμη, το κλείσιμο κάποιων περιοχών των περιοχών, δηλαδή όπου τα πιο ευάλωτα ήδη έχουν καλές ε, ευκαιρίες επιβίωσης, ε, να αποτελέσει λύση. Και όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, η μείωση της θνησιμότητας του ΕΦ φαίνεται να είναι απαραίτητο να είναι υψηλή. Δεν ξέρω ποια θα πρέπει να είναι η προθεσμία για τις μειώσεις αυτές. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανεί ε, όσο πιο σύντομα τόσο, το καλύτερο, διότι αν διατηρηθεί ψηλά το F τότε υπάρχει η πιθανότητα καταστροφή των αποθεμάτων, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουν όσοι ασχολούνται με τη διαχείρισή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Όχι, ωραία. Οπότε να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά και να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα που είναι και το πιο συγκεκριμένο και αφορά την αξιολόγηση του κανονισμού, των επιπτώσεων του κανονισμού και της εφαρμογής του στην Μεσόγειο. Θα δώσουμε τον λόγο λοιπόν στην Μονίκ Παριά που είναι διευθύντρια για την Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα στην DG ε, Mare και μετά θα συνεχίσουμε με τους διάφορους άλλους συγκεκριμένους μας προσκεκλημένους. Έχετε τον λόγο κυρία Παριά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η παρουσίασή μου θα γίνει σε δύο μέρη. Θα κάνω πρώτα μία εισαγωγή και μετά θα σας δείξουμε διαφάνειες με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που οργανώσατε αυτήν την πολύ επίκαιρη ακρόαση που πραγματοποιείται σε πολύ κρίσιμη στιγμή για την αλληλεία της Ευρώπης. Η θέση σε ισχύ του, της αναθεωρημένης πολιτικής πλησιάζει και είναι καλή η στιγμή αυτή να κοιτάξουμε το παρελθόν, να δούμε τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Και για να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την πολιτική για να ε, αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Όπως γνωρίζετε, η αλληλεία στην Μεσόγειο δεν ρυθμίζεται μόνο από τον βασικό κανονισμό για την κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά και από συγκεκριμένο κανονισμό για την Μεσόγειο που υιοθετήθηκε στο, στα τέλη του 2007 μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Με τον κανονισμό αυτό εισάγεται μία προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα διαχείρισης των, ε, της αλληλείας τους με την υποχρέωση να καθορίσουν ε, προγράμματα διαχείρισης ιδιαίτερα για την ε, αλληλεία που πραγματοποιείται με δίχτυα τράτας, ρήπους ε, βάρκα, ε, πεζότατε, κυκλωτικά δίχτυα και δράγες ε, στα εδαφικά ύδατα. Το σχέδιο δράση αποτελεί τρόπο για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένη της κακή κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο. Ο κανονισμό για τη Μεσόγειο περιέχει διατάξεις για την δημιουργία προστατευόμενων περιοχών και για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Υπάρχει ελάχιστο μέγεθος αλίας για κάποια ευάλωτα είδη, ελάχιστες αποστάσεις και βάθη για τον ε, εξοπλισμό της αλίας και άλλα τεχνικά μέτρα. Ο κανονισμός τέθηκε πλήρως σε ισχύ τον Ιούνιο του 2010. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού και ιδιαίτερα κατά τον καθορισμό των σχεδίων διαχείρισης. Παρά τη μεταβατική περίοδο δεν έχει οθετηθεί σχέδιο τον Ιούνιο του 2010. Έκτοτε όμως, χάρη στις κοινέ προσπάθειες των κρατών μελών και της Κομισιόν, η Κομισιόν έχει βελτιώσει την κατάσταση. Ο Φαμπρίς θα σας δώσει πιο καθαρή εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά να πω ότι τα δύο τρίτα του σχεδίου διαχείρισης του κανονισμού για τη Μεσόγειο έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό απέτησε μεγάλε επενδύσεις και για την διοίκηση των κρατών μελών και για τι υπηρεσίε τη Κομισιόν, αλλά πάντως εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Έχουν καταβληθεί επίσης προσπάθειες ε, να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που θα πρέπει να προστατευτούν, αλλά απομένει ακόμα δουλειά να γίνει στον τομέα αυτών. Να απαντήσω και στην ερώτηση του κυρίου Ρωμέβα. Προφανώς είναι πολύ νωρί να αξιολογήσει κανεί πόσο αποτελεσματικά τα σχέδια αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν την ε, ανισχυτικά κατάσταση για τα περισσότερα εμπορικά είδη. Υπάρχει υποχρέωση να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό το προβλέπει η μεταρρύθμιση. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρακολουθήσουν την εφαρμογή αυτήν πολύ προσεκτικά και να προχωρήσουν στην απαραίτητη προσαρμογή των σχεδίων αυτών για να καλυφθούν οι απαιτήσει. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, στην Μεσόγειο, που θα αφορά και την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και την περιφερειοποίηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Φαπρίτσιο που θα σας παρουσιάσει κάποιες διαφάνειες, τις οποίες βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσες για να σας δώσει μια εικόνα των πόσων σχεδίων διαχείρισης έχουν υιοθετηθεί, πού βρισκόμαστε ποια εξετάζονται ακόμα. Και επίσης για να σας δώσουμε μια επισκόπηση του τι καλύπτεται και όσον αφορά τις περιφέρειες και όσον αφορά τα αποθέματα που καλύπτονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, ναι, σας ακούμε. Thank you, Chair. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε η κυρία Πάρια, μπορούμε σήμερα να σας δώσουμε μια επισκόπηση των όσων έχουν πραγματοποιηθεί από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη Μεσόγειο και ιδιαίτερα του κανονισμού για τη Μεσόγειο, που είναι ο κανονισμός που υιοθετήθηκε το 2006 και τέθηκε σε ισχύ το 2007 και που καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη για να εφαρμοστούν οι κανόνες της κοινής αλληλευτικής πολιτικής στη Μεσόγειο. Αποφασίσαμε λοιπόν να σας δώσουμε μια εικόνα με βάση τρεις βασικές υποχρεώσεις, και τις οποίες επιλέξαμε, διότι θεωρήσαμε ότι είναι οι πιο σημαντικές. Αλλά βέβαια όσοι έχουν διαβάσει τον κανονισμό για τη Μεσόγειο γνωρίζουν ότι αυτά αποτελούν μόνο μέρος αυτού του πολύπλοκου νομοθετήματος. Να ξεκινήσουμε από τα σχέδια διαχείρισης. Κάτι που ήδη έχουμε εντοπίσει ως ε, βασικό στοιχείο. Προβλέπεται λοιπόν στο άρθρο 19 μέχρι το τέλος ε, του Δεκεμβρίου του 2007 να υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σε διάφορα είδη εξοπλισμού. Όπω είπε η κυρία Παριά, μέχρι το 2010 δεν είχε υιοθετηθεί τίποτα ακόμα από τα κράτη-μέλη. Τρία χρόνια αργότερα βρισκόμαστε σε θέση όπου συνολικά 27 σχέδια διαχείρισης έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη για τα πιο βασικά είδη εξοπλισμού για την αλληλεία. Δηλαδή για τις τράτες, για τα γρηγρή και για τους γρήπους βάρκας. Και εάν κοιτάξετε την κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, φέτος τον Μάιο είχαμε την ευκαιρία να πείσουμε τα μέλη του GFCM να υιοθετήσουν ένα σχέδιο διαχείρισης για το σύνολο της Αδριατικής. Σήμερα λοιπόν έχουμε 27 εθνικά σχέδια δράσης και ένα σε, εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει σχετικό έγγραφο που δίνει πολύ λεπτομερείς πληροφορίες σε σχετικά με αυτά τα σχέδια διαχείρισης. Αν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, βλέπουμε εδώ τα διάφορα σχέδια ε, διαχείρισης που έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη. Στην Κροατία έχουν αναλυθεί κάποια μέτρα πριν την προσχώρηση αλλά και μετά. Αλλά κατά τα άλλα, τα περισσότερα έχουν υιοθετήσει κάποια σχέδια, κάποια ετοιμάζονται ακόμα, κάποια υιοθετούνται, εγκρίνονται. Και η κατάσταση εξελίσσεται αρκετά γρήγορα. Η τελευταία συζήτηση που είχαμε με τα κράτη-μέλη ήταν ε, μετά του TCF το Νοέμβριο όπου εγκρίθηκαν κάποια σχέδια και από την επιστημονική κοινότητα. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα και όπως σας είπα εκτός από την Κροατία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μέσα στα προηγούμενα 3,5 χρόνια έχει πραγματοποιηθεί πολλή δουλειά για να εφαρμοστεί αυτή η υποχρέωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία αξιολογούνται ή αναθεωρούνται Κάνουν πολλή δουλειά τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουν σχέδια τα οποία να βασίζονται στις τελευταίες επιστημονικές πληροφορίες. Σίγουρα μπορούμε να επανέλθουμε στα σχέδια αυτά. Και όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή, βλέπετε εδώ μια εικόνα, ένα στιγμιότυπο της κάλυψης των σχεδίων διαχείρισης για τα διάφορα είδη εξοπλισμού. Βλέπετε λοιπόν τη γεωγραφική κάλυψη για τις στράτες, εδώ για τα γρηγρή και τέλος για τους γρήπους βάρκας. Βλέπετε ότι υπάρχει ανεπαρκής κάλυψη σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτά είναι τα σχέδια που ήδη έχουν υιοθετηθεί. Δεν είναι αυτά που αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται ή αναθεωρούνται. Εάν συνδυάσουμε τα τρία είδη εξοπλισμού, βλέπετε πού βρισκόμαστε σήμερα. Βλέπετε έτσι την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2010, τρία χρόνια μετά την έγκριση του κανονισμού για τη Μεσόγειο, δεν έχουν που δεν είχαν υιοθετηθεί σχέδια από τα κράτη-μέλη. Βλέπετε λοιπόν τώρα τα σχέδια που έχουν εγκριθεί με βάση το νομικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε. Αυτή η εικόνα δείχνει που βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά την κάλυψη για την διαχείριση της ελίας. Υπολογίζουμε ότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, απομένει πολλή δουλειά να γίνει για να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα ενισχυτική κατάσταση των αποθεμάτων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες, όχι μόνο για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, αλλά και για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συνέχεια που θα δοθεί. Οι απαραίτητες προσαρμογές θα πρέπει να γίνονται με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες. Με λίγα λόγια, το 2010 δεν υπήρχε τίποτα. Έχει γίνει πολλή δουλειά στο μεταξύ, έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για να καλύψουμε την αλία και να μπορούμε να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες αλίας στη Μεσόγειο. Οι περισσότερες αξιολογήσεις της ΣΤΕΚ γίνανε στο διάστημα 2010-2012, κατά την έναρξη δηλαδή της εφαρμογής αυτής της υποχρέωσης. Η σχέση λοιπόν ανάμεσα στην έγκριση και την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης ε, πρέπει να αξιολογηθεί για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τα κατάλληλα μέτρα για να καλύψουμε αυτή την υποχρέωση. Η δεύτερη σημαντική υποχρέωση που θελήσαμε να καλύψουμε είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να δημιουργήσουν περιοχές προστατευμένες. Αυτό συνδέεται με την ύπαρξη σχεδίων διαχείρισης για την παρακολούθηση της ε, αλλιευτικής δραστηριότητας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στον σχετικό κανονισμό. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε μέχρι το τέλος του 2007 να υποβάλουν στοιχεία για τις προστατευόμενες περιοχές που ήδη είχαν δημιουργηθεί και να συνεχίσουν να δημιουργούν τέτοιε με πιο συστηματικό τρόπο μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2007. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Κάποιες από αυτές τις προστατευόμενες περιοχές συνδέονται με την εφαρμογή άλλων νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες συνδέονται με σχέδιο διαχείρισης, κάποιες συνδέονται με άλλου τύπου υποχρεώσεις. Σήμερα είχαμε μια κάποια επισκόπηση του πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά την κάλυψη αυτής της υποχρέωσης. Εκτός από την Κροατία, για την οποία ακόμα γίνεται η επαλήθευση, γνωρίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν επιβεβαιώσει απέναντι στην Κομισιόν ότι έχουν δημιουργήσει προστατευόμενες περιοχές. Είναι πιο δύσκολο να σας παρουσιάσουμε την γεωγραφική κάλυψη, διότι δεν είναι όλες οι περιοχές όμοιες, δεν καλύπτουν δύο τύπου υποχρέωση, ωστόσο γνωρίζουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία θα συνεχίσει να είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή του νέου βασικού κανονισμού, του οποίου η εφαρμογή θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Το τρίτο στοιχείο που συνδέεται με την ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων και προστασίας κάποιων ειδών είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να έχουν σωστή χαρτογράφηση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Υπάρχουν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε ευαίσθητες περιοχές δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει σαφής εικόνα εάν δεν υπάρχει σωστή χαρτογράφηση. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση σίγουρα στη Μεσόγειο και έχει δημιουργήσει δυσκολίες όσον αφορά να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Πολλά κρατημέλη έχουν πληρώσει αυτή την υποχρέωση είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνται δραστηριότητες πάνω σε οικοσυστήματα που θα πρέπει να προστατευτούν περαιτέρω και που θα πρέπει να αξιολογηθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν μέτρα διαχείρισης, τα οποία είχαν ληφθεί από τα κράτη-μέλη ήδη πριν τη θέση σε ισχύ του κανονισμού για τη Μεσόγειο, για να προστατευτούν αυτά τα οικοσυστήματα που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες αλίας. Αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά τα λεγόμενα Posidonia Beds, τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο στον κανονισμό για την Μεσόγειο, Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να δούμε πού βρισκόμαστε. Γνωρίζουμε σήμερα ότι απομένει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει. Η δουλειά συνεχίζεται. Συνοψίζοντας λοιπόν Υπάρχουν ε, οι συμφωνίε εταιρική σχέση στον τομέα τη αλληλεία, υπάρχουν και άλλα νομοθετήματα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι αποκλειστικά αλλιευτικό, ούτε συνδέεται αποκλειστικά με τη Μεσόγειο. Έχει να κάνει με πολλές άλλες υποχρεώσεις και υπάρχει προσπάθεια να Υπάρχουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης σε διάφορους τομείς, ε, καθώς και εθνικά σχέδια διαχείρισης. Ε, στη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική, η προστασία των οικοσυστημάτων θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Και πολύ σύντομα, για να ολοκληρώσω αυτή την ε, σύντομη παρουσίαση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει σημειωθεί πολύ πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η πρόοδος είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο δεν βρισκόμαστε ακόμα σε θέση να πούμε ότι έχουμε πετύχει τον στόχο μας, ε, το αντίθετο θα έλεγα, και θα ήθελα ε, να αναφερθώ και στην ε, παρουσίαση που έγινε πριν σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων. Συνειδητοποιήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στις εθνικές διοικήσεις που εφαρμόζουν τον κανονισμό, αυτές που εκπονούν τα σχέδια διαχείριση ε, και άλλου ενδιαφέρομένου. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην εξετάζουμε τον κανονισμό περί Μεσογείου ή την κοινή αλληλευτική πολιτική στη Μεσόγειο ως απομονωμένο θέμα και στη Μεσόγειο υπάρχουν πολλά μοιρασμένα αποθέματα όσον αφορά την περιοχή, όσον αφορά την αλληλεία Έχουμε όμως και πολλά αποθέματα που μοιραζόμαστε με μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντονισμό των μέτρων διαχείρισης και των κανόνων είναι απαραίτητος για να πετύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για τα αποθέματα αυτά. Αυτές λοιπόν είναι οι προκλήσεις και θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειε ε, του επόμενου μήνε και τα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνέ επίπεδο. Σα ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε κάτι να πείτε ακόμα, κυρία Παριά, από πλευρά τη Κομισιόν, πριν να δώσω το λόγο στου ε, βουλευτέ. Όχι, ωραία. Οπότε ξεκινάμε τον ε, γύρο ερωταπαντήσεων με του ε, ευρωβουλευτέ. Η κυρία Φράγα, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Κομισιόν. Εγώ, καταρχήν, θα ήθελα να ρωτήσω Πότε προβλέπει να την υποβολή μεταρρύθμιση αυτού του κανονισμού, τροπολογία ε, αυτού του κανονισμού, για να προσαρμοστεί στη νέα και κοινή αλληλευτική πολιτική. Ε, είναι όντω αλήθεια ότι δεν εφαρμόζεται στη Μεσόγειο το θέμα των ε, εκφορτώσεων ή απορρίψεων. Ήθελα επίσης να ρωτήσω κάτι για το άρθρο 9, δηλαδή το μήνυμο μέγεθος για τα μάτια των δικτυών. Ε, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εσείς λέτε ως τελική κοσυμπέρασμα ότι αυτό το άρθρο δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Όμως έπρεπε αυτό να έχει εφαρμοστεί πλήρως από το 2010. Και εσείς λέτε τώρα πως δεν έχει πλήρως εφαρμοστεί. τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και έπειτα μου τράβηξε την προσοχή ότι ένα κράτος μέλος όπως η Γαλλία το με... οι μισές ε, τράτες βυθού δεν συμμορφώνονται προς αυτήν την... Ε, σε αυτό το κανονισμό. 20 χιλιοστά είναι το μέγεθος των ματιών, λιγότερο από το μισό δηλαδή που είναι υποχρεωτικό. Ε, πώς καταλα... Δεν καταλαβαίνω πώς το δέχεται αυτό η Κομισιόν, ενώ στο άρθρο 9 δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση από αυτό το μέγεθος. Επιπλέον, μου τραβήξε την προσοχή αυτό που είπατε πως στην πράξη Είσατε, δέχεστε μάλλον την αλλαγή στις 25, στις 25 μάτια. Δεν ταιριάζουν αυτές, ε, αυτά τα νούμερα με το σύνολο των ε, γρηγρή και τρατών που υπάρχουν στο Μεσόγειο. Γιατί ξέρουμε και ότι στον προηγούμενο κανονισμό υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα νούμερα για το μέγεθος των ματιών. Τέλος, να σας ρωτήσω το εξής. Το άρθρο 9 προβλέπεται η δυνατότητα να είναι 40 χιλιοστά το μάτι ή μέχρι 50 χιλιοστά όταν υπάρχει δικαιολογία, όταν υπάρχει αιτολόγηση. Τώρα, Ε, μόνο τα 90 ε, σκάφη που κυκλοφορούν είναι αυτά που, κυκλοφορούν τα, που χρησιμοποιούν τα τετράγωνα μάτια δικτυών ενώ τα υπόλοιπα 1430 χρησιμοποιούν ε, τα ρομβοειδή δίχτυα ε, δεν θα πρέπει αυτό να το αλλάξουμε ώστε, γιατί είναι πιο φτηνά, γιατί είναι πιο ανθεκτικά κτλ. κτλ. Ξέρουμε γιατί. Αλλά εν πάση περιπτώσει αφού ο κανονισμός λέει κάτι άλλο ε, ε δεν θα πρέπει να, μην το, να, το, να το καταργήσουμε, να μην ισχύει πλέον ως εξαίρεση γιατί το 75% των σκαφών έχουν αλλάξει σε αυτό το είδος ε, ματιού το ρομβοϊδές. Σας ευχαριστούμε κυρία Φράγα. Ο κύριος Άγνιου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές, για αυτές τις πολύ καλές παρουσιάσεις. Είναι απελπιστική η κατάσταση στην Μεσόγειο από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι κατάλαβα το 95% των ειδών απειλούνται και για να διορθωθεί η κατάσταση θα πρέπει να μειωθεί στο μισό η αλληλευτική προσπάθεια. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και ναι, η κατανόηση του προβλήματος ε, είναι η μισή δουλειά, αλλά όπως είπατε, η εφαρμογή και η επιβολή του νόμου ε, είναι η υπόλοιπη δουλειά. Είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο. Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή και δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα εξαντλήσουμε τα αποθέματα στη Μεσόγειο ή θα πρέπει να παραμένουν στα λιμάνια το μισό των αλλιευτικών σκαφών για πάντα. Κάτι που ε, θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες για την επιβολή του νόμου. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν γι' αυτό. Η Μεσόγειος είναι μια λίμνη ουσιαστικά με μια μικρή πρόσβαση τον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι ομοιογενής επιτροπή ε, περιοχή και δεν είναι πολύ εύκολο να ελέγξουμε όλον το στόλο, διότι υπάρχει και ο, ο στόλος της Βορείου Αφρικής. Δεν αναφέρθηκε η αλληλευτική προσπάθεια αυτού του στόλου. Μπορείτε να μας πείτε αν εκείνοι υπεραλλιεύουν το δικό τους μισό. Και ακόμα και αν ε, και τα 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Μεσόγειο Εάν συμμορφωθούν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αναιρεθεί τελείω από την αλληλευτική προσπάθεια των χωρών της Βόρειας Αφρικής. Ευχαριστώ κύριε Άγγλιο. Η κυρία Λοβέν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Νιώθω κάποια αισιοδοξία όταν βλέπω τα νέα σχέδια διαχείρισης ε, τα οποία επιτέλους εφαρμόζονται τα τελευταία τρία χρόνια. Νιώθω όμως ε, και κάποια οργή όταν ακούω ότι κανένα από τα κράτη-μέλη της Μεσογείου δεν είχαν εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης μέχρι το 2010, παρότι έπρεπε να το έχουν κάνει αυτό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2007. Η Κομισιόν φαντάζομαι θα είναι πολύ ευγενική για να μας πει γιατί, αλλά μήπως μπορείτε να μας πείτε η Κομισιόν τι προσπάθησε να κάνει για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι. Και αν υπήρξαν κυρώσεις εις βάρος των κρατών μελών για το λόγο ότι δεν προσπάθησαν καν να δημιουργήσουν την νομοθεσία στην οποία ήδη είχαν συμφωνήσει το 2006. Δεν μιλάμε για ξένες δυνάμεις που συμφώνησαν πάνω στην νομοθεσία αυτή. Τα ίδια τα κράτη-μέλη συμφώνησαν και δεν έκαναν τίποτα. Για μένα είναι τρομερό ότι υπήρχε αυτή η κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων. Τουλάχιστον τώρα έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος και αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι πρώτη φορά που ακούω παρουσίαση για τη Μεσόγειο στην οποία να ακούμε για πρόοδο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ θετικό. Για πρώτη φορά λοιπόν ακούμε κάποιες απαντήσεις, ακούμε ότι υπάρχουν σχέδια διαχείρισης για τα διάφορα είδη αλληλείας. Ερώτηση, πόσα ακόμα σχέδια απομένουν να προετοιμαστούν κατά τη γνώμη της Κομισιόν. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόντοστ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησαν η κυρία Φράγα και η κυρία Λεβίν. Θα ήθελα να πω ότι βρίσκω τρομερό ότι από το 2006 μέχρι το 2013 έχουμε φτάσει σχεδόν στην πρωτοχρονιά, σχεδόν 2014 έχουμε. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι λοιπόν πολύ πενιχρά τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το 2007 έπρεπε ήδη να έχουν καθοριστεί οι προστατευόμενες περιοχές και ακούμε ότι το 95% των αποθεμάτων συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο υπεραλίας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει ο νέος κανονισμός, ο νέος βασικός κανονισμός ε, για να δοθεί τέλος στην κατάσταση αυτή. Συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Πολεμάμε συνέχεια με το Συμβούλιο Σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης, ε, το Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν πρέπει να συναποφασίζουμε. Εγώ βρίσκω καταστροφική και την κατάσταση στη Μεσόγειο. Αυτό δεν θα έπρεπε να αρκεί ώστε να συμμορφωθεί το Συμβούλιο. Και η Κομισιόν στο μέλλον τι θέση θα κρατήσει. Είπατε ότι θα πρέπει να γίνει ο ε, να υπάρχει έλεγχος, παρακολούθηση. Είναι όμως μακρύ το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, είναι κάτι που απαιτεί χρόνο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και όχι πριν, όσον αφορά την Μεσόγειο, και θα πρέπει να αναπτύξουμε μέσα ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα διότι αλλιώ θα καταστραφούν τελείω τα αποθέματα εκεί και αυτό δεν είναι προ συμφέρον των αλλιέων που εξαρτώνται από την αλληλεία. Από το 2006 μέχρι σχεδόν το 2014, 8 χρόνια, δεν έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Βρίσκω πενιχρά τα αποτελέσματα, δεν θέλω να επιτεθώ σε εσά προσωπικά, αλλά βρίσκω ότι είναι πενιχρά τα αποτελέσματα. Έχω μείνει άφωνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Να κάνω κι εγώ παρατηρήσεις προς την ίδια κατεύθυνση, δύο-τρεις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η στην διαδικασία υιοθέτηση τη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική έχουμε ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο την Μεσόγειο και αυτό πληρώνουμε τώρα τρόπον την Υπάρχουν ιδιαιτερότητε στη Μεσόγειο και κάποια από τα θέματα κλειδιά δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς. Και τώρα αντιμετωπίζουμε την ανάγκη να έχουμε νέα μέσα, νέα εργαλεία. Κάποια πειράματα μπορεί να φανούν χρήσιμα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην συνδιαχείριση. Που θα αποτελέσει λύση σε κάποια από τα σύνθετα αποθέματα. Κάποια αποθέματα είναι, έχουν απλή σύνθεση, οπότε είναι πιο εύκολο να ασχοληθούμε με αυτά. Αλλά τι γίνεται όσον αφορά τη συνδιαχείριση, όπου συμμετέχουν πολλοί παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την διαχείριση κάποιων αποθεμάτων. Γνωρίζω ότι στη Μεσόγειο συμβαίνει αυτό. Δεύτερη ερώτηση αφορά όχι μόνο την χαρτογράφηση των ε, θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών, αλλά και των αποθεμάτων και των ζωνών προστατευμένης αλληλείας. Πώς σχεδιάζουμε να συνδέσουμε όλες αυτές τις διάφορες περιοχές οι οποίες αποτελούν και μέρος του όλου χάρτη και θα πρέπει να τις δούμε σε συνδυασμό με την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, δεν αρκεί μόνο η χαρτογράφηση των προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει σίγουρα να γνωρίσουμε πού βρίσκονται οι περιοχές αυτές, αλλά το ανέφεραν αυτό και οι άλλοι συνάδελφοί μου. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν πολιτική βούληση, ώστε να διαθέσουν πόρους και χρήματα, ώστε οι προστατευόμενες περιοχές αυτές να προστατευτούν σωστά. Τι γίνεται λοιπόν στον τομέα αυτόν. και πώς γίνεται αυτό στο πλαίσιο της εφαρμογής ε, της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, ε, αλλά και του EMFF, του Ταμείου για την Αλία και τη Θάλασσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλη παρέμβαση από άλλον ε, Ευρωβουλευτή, οπότε θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Παρακαλώ, κυρία Παριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πριν απαντήσω για κάθε ερώτηση, θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν έκαναν τίποτα πριν από το 2010. Έτσι έχει η κατάσταση μου. Αλλά ίσως θα έπρεπε σε πιο θετικό πνεύμα να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που τα κράτη-μέλη έχουν φτιάξει με πολλές δυσκολίες και φυσικά όρα που έχουν από την τελειότητα, πάντως έχουν φτιάξει διαχειριστικά ε, πλάνα για την αλληλεία τους. Και όπως σας λέω, δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ πριν. Μας πήρε όντως τρία χρόνια πολύ σκληρές προσπάθειες. Έχουμε λοιπόν 39 διαχειριστικά πλάνα μαζί με τα κράτη-μέλη. Σχεδόν κάθε μήνα είχαμε συνεδριάσει μαζί τους τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτά τα σχέδια. Δεν ξέρω πόσες πολλές διαδικασίες έχουμε χάσει Κάθε κράτος μέλος έχει, είναι σε διαδικασία διαφοράς, παραβάσεις, λόγω του ότι δεν εφάρμοσαν τον κανονισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι των διαχειριστικών σχεδίων. Κάναμε ελέγχους και έτσι απαντώ στο θέμα της, ε, του σεβασμού της δικής μας αποστολής. Κάνουμε τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους ελεγκτικές αποστολές στις περισσότερες χώρες και κάθε παράβαση ε, καταγράφεται, τη παρακολουθούμε και αν χρειάζεται προβαίνουμε και σε διαδικασίες κατά παράβαση δεν ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Η ίδια διαδικασία ισχύει για όλους. Δεν επιτρέπουμε κάτι σε μια χώρα το οποίο παγορεύουμε σε κάποια άλλη. Ο κανόνας λοιπόν για το μέγεθος των ματιών, για τα... τις στράτες ισχύει για όλους. Και ακόμα συζητάμε με κάποια κρατημέλη για την εφαρμογή και το σεβασμό του μεγέθους των ματιών για τις στράτες. Οι συνάδελφοι θα μιλήσουν για τις ιδιαιτερότητες του μεγέθους των, των ματιών, αλλά θα ήθελα να πω ότι τα μεγέθη ματιών που αναφέρονται στον κανονισμό είναι τα μικρότερα και είναι μάλλον το ελάχιστο. Ε, λέμε, μάλλον ο κανονισμός λέει τουλάχιστον αυτό πρέπει να το σεβαστούν. Αν τα κάτι θέλουν μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. The situation is worrying and we are fully aware of that. Τώρα, η κατάσταση είναι όντως ε, επικίνδυνη, το γνωρίζουμε και γι' αυτό ακριβώς και ήμασταν και τόσο αυστηροί να συσταθούν αυτά τα σχέδια, τουλάχιστον να αποτελέσουν μια βάση. Πιθανότητα δεν θα αρκέσουν για να ανταποκριθούμε στις ε, πολύ ε, σημαντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, αλλά τουλάχιστον είναι μια βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε. Και όπως έχω πει και παλιότερα, αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Ο γαλάζιος τόνος εφαρμογή των ε, ελέγχων για τις στραταληπτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητές μας. Ε, και όπως έχω πει και παλιότερα και το είπατε και αρκετοί από εσά και σωστά, η Μεσόγειος είναι μια λίμνη στην ουσία. Ακόμα και αν τα κρατημέλη σεβαστούν τον κανονισμό, την ομοθέσια, δεν θα αντιμετωπιστεί πλήρως η κατάσταση των ε, αποθεμάτων και γι' αυτό αρχίσαμε ταυτόχρονα τα τελευταία τρία χρόνια μια μεγάλη επισκόπηση της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας για τη Μεσόγειο, γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη Μεσόγειο εάν δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες. Και όχι μόνο οι Αφρικανικές, είναι και η Τουρκία, είναι δηλαδή και η ανατολική πλευρά των όχθεων της Μεσογείου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μέτρα αλλά και πάλι με την γενική επισκόπηση της GFCM που βασικά γείται αυτή η ένωση γιατί είναι ο κύριος εταίρος. Έχουμε σχετικά ανοιχτή υποστήριξη από την Τουρκία. Καταφέραμε πέρσι για πρώτη φορά να έχουμε ένα σχέδιο διαχειριστικό για την GFC, για την Αδριατική, για τα μικρά πελαγικά είδη που είναι από αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο. Ήδη λοιπόν αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Το δέχομαι ότι πρέπει να γίνουν πολλά και ότι είμαστε μόνο στην αρχή μιας διαδικασίας. Το αναγνωρίζω ότι αυτή η διαδικασία έπρεπε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Πρέπει όλα αυτά λοιπόν να τα παρακολουθούμε και όπως είπε και ο κύριος Ρωμέβα, πρέπει να εφαρμόσουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής στη Μεσόγειο γιατί και η κυρία Φράγα ρώτησε σχετικά με αυτό, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις ε, εκφόρτωσης, την, τον MSY στη Μεσόγειο όπως και σε άλλες περιοχές της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει αυτό την επόμενη χρονιά για τα μικρά απαλλαγικά είδη και η φόρτωση μας υποχρεώνει μέχρι το 2015 οπότε θα εισαχθεί αυτό τον επόμενο χρόνο όπως και σε άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Μεσογείου και επίσης αρχίσαμε να δουλεύουμε με τα κρατημέλη και με τις, ε, με την ε, ενώσει των αλλιέων. Θα ακούσουμε και τον κύριο Μπομφίλιο αργότερα που την, τις εκπροσωπεί εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση. Έγινε και, και πέρσι αυτό με την αλλαγή της ε, προεδρίας στο RACMED και θα εφαρμοστούν αυτά τα, τα μέτρα. Εάν χρειαστεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός της Μεσογείου, θα το δούμε, γιατί κατά τη γνώμη μα είναι πολύ νωρί για να αλλάξουμε κάτι το οποίο δεν έχει στην ουσία εφαρμοστεί Πλήρω μέχρι τώρα. Δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να το εξετάζουμε στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινή ελευτικής πολιτικής της ε, μεταρρύθμισης αυτής και επί τη βάση επίσης της αξιολόγησης των όσων έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ε, και όπως είπα από την αρχή, όταν το να αξιολογήσουμε κάτι πάση πριν από ένα-δύο χρόνια, ούτε καν, είναι πολύ νωρίς κατά τη γνώμη μου. Μέτρα συν διαχείρισης. Έχουμε μία περιφέρεια και μία αλληλεία στην Ισπανία που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία διαχείριση, Είναι κάτι το οποίο προωθούμε, το βαθμολογούμε επίσης και το προωθούμε και προς τις άλλες χώρες ως έναν τρόπο για να γίνει καλύτερη διαχείριση των αλλιευμάτων στην Μεσόγειο και είναι θετική η εμπειρία που αποκομίζουμε. Για τη χαρτογράφηση των διαφόρων ε, περιοχών αλίευσης. Δουλεύουμε γι' αυτό τους επόμενους μήνες. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω για την ώρα, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς μαζί σας. Βασική μας, ε, βασικός μας στόχος και ε, πίεση υπήρχε για το θέμα των σχεδίων διαχείρισης και γι' αυτό τα άλλα τα είχαμε κάπως παραμελήσει. Τώρα θα πιέσουμε περισσότερο και γι' αυτά. Τώρα, Πρέπει να χρηματοδοτηθούν ε, οι περιοχές ε, Natura 2000, ε, οι προστατευόμενες περιοχές αλληλείας και όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στους ορισμούς και, και, τα χρησιμοποιούμε στη σύσταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών, τους ορισμούς αυτούς, αλλά πραγματικά θα εκτιμούσαμε τη δική σας στήριξη στην επαφή με τα κράτη-μέλη, ώστε να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή αυτών των σχεδίων σχεδίων όταν πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, και πιθανότατα θα χρειαστεί και να προσαρμοστούν για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τα MSY στα επόμενα χρόνια. και να λάβουμε υπόψη και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τη μεταρρυθμισμένη κοινή ελευτική πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θέλει κανείς να πει κάτι εξ ονόματος της Επιτροπής. Άλλος, όχι. Η κυρία Φράγα. Εγώ ακούω πάρα πολύ προσεκτικά τα όσα λέει η κυρία Παριάτη και μένει μια ερώτηση που είναι σε κρεμότητα στην οποία δεν μου απάντησε και είναι το θέμα των τρατών στο ένα κράτος μέλος συγκεκριμένο που χρησιμοποιεί μάτια 20 χιλιοστών. Θέλω να γνωρίζω γιατί και πώς επιτρέπει η Κομισιόν το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί κάποιο κράτος να έχει πιο μεγάλα μάτια από αυτό που προβλέπει ο κανονισμός, αλλά όχι πιο μικρά. Κάνει κάτι η Κομισιόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ε, αυτή ήταν η ερώτησή μου και δεν έλαβα απάντηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση, η κυρία Παριά. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε μάλλον δεν ήμουν σαφής, αλλά δεν υπάρχει εξαίρεση για το μέγεθος των ματιών. Αν κάποιο κράτος μέλος εξακολουθεί να επιτρέπει τράτες με μάτια δικτυών που δεν συμμορφούνται προς τον κανονισμό της Μεσογείου, φυσικά θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και ακόμα γίνονται συζητήσεις με ένα συγκεκριμένο κράτος ε, για αυτό το θέμα και γι' αυτό και δεν έχει οθετηθεί και το σχέδιο του. Μάλιστα. Bien. No hay ninguna otra cuestión. Μάλιστα, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ε, περνάμε στο δεύτερο τμήμα αυτού του δεύτερου τμήματος. κύριε Άγνιου, ναι, συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές, ότι, ναι, αυτό θα έλεγε ο Άγνιου, αλλά έχοντα ακούσει αυτά που μόλις είπε η Κομισιόν, ελπίζουν να λάβουν χρήματα για να βελτιωθεί η καταστροφική κατάσταση αυτή στην Μεσόγειο και ποιος θα τα δώσει αυτά τα χρήματα, ο Βρετανός φορολογούμενος ε, που δεν έχει καμία σχέση με το Μεσόγειο. τουλάχιστον γελάτε. Σας ευχαριστώ κύριε Άγνιου. Πάντα μας διασκεδάζουν τα σχόλιά σας, ναι. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα με τρεις παρεμβάσεις, τρεις εισηγήσει, μία μετά την άλλη, όμως δεν θα κάνουμε ερωταπαντήσεις μετά από κάθε εισήγηση. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι τρεις και μετά θα τις κάνουμε ερωτήσεις. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Τζαμπάολο Μπομφίλιο, που είναι πρόεδρος του Ένωσης των Ιταλικών Συνεταιρισμών Αλληλείας. Κύριε Μπονφίλιο, έχετε το λόγο. Scusate. Grazie Presidente, grazie per l'invito, grazie per questa audizione. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ακρόαση που διοργανώσατε. Μάλιστα εδώ και χρόνια ελπίζαμε ότι θα εξεταστεί εκ νέου αυτός ο κανονισμός γιατί ε, Όχι ότι θα γίνουν τίποτα τρομερές αλλαγές, αλλά γιατί κατά τη γνώμη μας όλα αυτά μπορούν να επαληθευθούν ε, και η λειτουργικότητά τους να εξολογηθεί και να βελτιωθεί. Και εδώ μιλώ με βάση την, ως εκπρόσωπος μάλλον της Ένωσης των Ιταλικών Συντερισμών Αλλιέων και θα είμαι πιο μεροληπτικός ε, από ότι όταν ε, μιλώ ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αλλιέων της Μεσογείου, ως εκπρόσωπος λοιπόν των αλλιέων θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον αντίκτυπο όχι μόνο στα ψάρια αλλά και στους αλλιείς, στην οικονομία των επιχειρήσεων, στη ζωή ολόκληρου του τομέα. Όπως λοιπόν ήδη αναφέρθηκε, Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006 μετά από μια μακρά διαδικασία κριτικών, ε, οξέων επικρίσεων, ε, προσπαθειών τροποποίησης και ούτω καθεξής. Άρχισε λοιπόν, εγκρίθηκε το 2006 και το Μάρτιο του 2007 άρχισε η εφαρμογή του χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερα τραύματα ή ε, ζημιές. Θα πρέπει αμέσω να πούμε ότι στην πράξη ε, είναι ένας κανονισμός που περιλαμβάνει πολλά τεχνικά μέτρα, πολλά ήδη αναφέρθηκαν, ε, τα δίχτυα, ε, τα μάτια των διχτυών, η απόσταση από τις ακτές, τεχνικές λεπτομέρειες δηλαδή των, της δραστηριότητα. δραστηριότητας και έπειτα υπάρχει και ένα μέγα τμήμα διαχειριστικό που είναι ακριβώς το, τα σχέδια τα διαχειριστικά για τα οποία ακούσαμε μόλις από την Επιτροπή. Όταν άρχισε λοιπόν η λειτουργία του, στην ορχία ε, άρχισε να ισχύει χωρίς προβλήματα γιατί τότε είχαν ε, αρχίσει ε, οι, οι ρυθμίσεις εκείνες τότε και υπήρχε το άρθρο το οποίο προέβλεπε μεταβατικές εξαιρέσεις και οι βασικές τεχνική, οι βασικοί μάλλον τεχνικοί κανόνες και αναφέρομαι στις ε, αξίες για απόσταση από τις ακτές και τη μήνυμα ε, μέγεθος ματιών για τις, ε, τα παρασυρώμενα δίχτυα. Στην ουσία αυτά όλα άρχισαν να ισχύουν οριστικό το 2010, τρία χρόνια αργότερα. Ήταν ένας κανονισμός δηλαδή ο οποίος άρχισε να ισχύει τουλάχιστον από τις τεχνικές του πλευρές σε δύο φάσεις το Μάρτιο του 2007 αμέσως ε, τα όρια για τις εκφορτώσεις άρθρο 15 και στη συνέχεια μια ολόκληρη σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών για τους αληφτικούς εξοπλισμούς που απαριθμώνται στα παραρτήματα 1 και 2 που αναφέρονται και τα άρθρα τα αντίστοιχα του κανονισμού. Ενώ όσον αφορά τα υπόλοιπα τεχνικά μέτρα τα οποία εγώ όρισα ως πιο σημαντικά για τις ελευτικές δραστηριότητες είναι εκείνα τα οποία είναι καταγεγραμμένα και πολύ θα το θυμάστε. Εκεί είδαμε διαμαρτυρίες, εντάσεις σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά λιμάνια και αλληλευτικές περιοχές. Ήταν τα δύο μέτρα που αφορούσαν το μήνυμο μέγεθος ματιών για τα παρασυρώμενα δίχτυα, τις αποστάσεις και τα βάθη για τη χρήση των ε, αλληλευτικών εξοπλισμών λοιπόν που άρχισαν να ισχύουν στις 31 Μαΐου του 2010. Στη συνέχεια όσον αφορά τα μήνυμα μεγέθη και εκεί υπήρχαν κάποιες ε, ανοχές, ε, ας πούμε το υπομέγεθος ε, του κάθε ε, ματιού έγινε δεκτό μέχρι 15% απόσταση μέχρι το τέλος του 2008. Δηλαδή υπήρξε μια σταδιακή ε, κατάργηση και προσαρμογή στον κανονισμό. Τώρα, αυτό που ήταν τελικά μια κίνηση που για όλους θα έπρεπε να είναι το 2007 και τελικά έγινε το 2010, εξηγείται έτσι και θυμίζω ότι αυτό το πρόβλημα των σχεδίων των διαχειριστικών του κανονισμού αυτού ήταν μια πτυχή η οποία κατά κάποιο τρόπο ε, ερχόταν και εφαπτόταν στο πλάνο διαχείρισης για την αλληλεία. Υπήρχαν δύο ειδών δηλαδή διαχειριστικά σχέδια. Το με, η μεσογειακή, ο μεσογειακός κανονισμός ζητούσε ε, τις ε, υδραυλικές ε, τράτες ε, ε, και ούτω καθεξής, ενώ και, αφορούσε το κάθε σύστημα. Ενώ τα σχέδια αλίες του, του Ταμείου αλίες, στην ουσία αφορούσαν το σύνολο των ελευτικών δραστηριοτήτων του, του GSA για το σύνολο της Μεσογείου όπως το είδαμε προηγουμένως. Και αυτή η επικάλυψη δεν βοήθησε στην, ε, στην εκκίνηση όλων αυτών των διαχειριστικών σχεδίων και οδήγησε σε μια κάποια ομολογουμένως καθυστέρηση. Τώρα, ε, κάποιοι είπαν ότι αν σκεφτούμε μια εφταετία και ακούμε να λέγεται πως το 95% ε, είναι υπεραλλιευόμενα ήδη, ε, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και εκείνη η παρουσίαση του Όσιο δεν μας κάνει και πολύ αισιόδοξου. Γιατί μιλάτε για το 55% των 50 στόκ, των 50 αποθεμάτων που αξιολογήθηκαν, ενώ στη Μεσόγειο υπάρχουν εκατοντάδες εκατοντάδων ήδη, ε, αν και βέβαια μπορεί στην ουσία να είναι η ίδια κατάσταση και για τα υπόλοιπα στόκ, αλλά μιλάμε για μια, ένα πρώτο, μια πρώτη ομάδα αξιολογήσεων. Φτάσαμε σε 40-50 αποθέματα που αξιολογήθηκαν και από αυτά το 95% είναι υπερελευόμενα. Αν όμως θεωρήσουμε ότι πολλά τεχνικά μέτρα έχουν αρχίσει να ισχύουν από το 2007, ενώ άλλα το 2010, τα διαχειριστικά σχέδια τώρα ξεκινάνε στην ουσία, σε σχέση με εκείνα τα στοιχεία τα ερευνητικά, τα, τη μέτρηση δηλαδή της ε, Εκμετάλλευση θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα γιατί δεν πάει καλά. Σε αυτό υπάρχουν ε, διαφορετικέ και αποκλίνουσες απόψεις. Αφήνονται όλα αυτά μόνο στην καθυστέρηση τη κατάθεση των διαχειριστικών σχεδίων που ξεκίνησαν το 2010 και οι επιστήμονε μα λένε ότι χρειάζονται τουλάχιστον τρία χρόνια για να, αξιολογηθούν, ε, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπο, ενώ εμεί πρέπει από τον επόμενο χρόνο να αρχίσουμε να βλέπουμε μια κάποια τάση εκεί δηλαδή που λειτουργήσαν τα σχέδια και που όχι έπειτα αν είναι ανεπαρκή και αναποτελεσματικά αυτά τα σχέδια θα το δούμε μετά από τρία χρόνια από την πραγματική τους εφαρμογή. Ίσως να πρόκειται για ανεπάρκεια των τεχνικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα που ίσως και κάποια να είναι λάθος ή θα μπορεί να οφείλεται σε μια ελλειπή εφαρμογή γενικευμένη. Αλλά αυτό θα σημαίνει πλήρη έλλειψη ελέγχου και αυτό μπορεί να αληθεύει μέχρι κάποιο σημείο, όπως είπε η Κομισιόν. Εγώ μπορώ να σας πω για κάποια ε, κατηγορίες υπάρχουν, ε, γίνονται έλεγχοι, γίνονται, υπάρχουν διαδικασίες κατά παράβαση και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα ελέγχου, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, ας δούμε για την κατηγορία και για τις ε, ε, συνεταιρισμούς αλίες, να δούμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις. Καταρχήν, μείωση του εισαλίευσης και σε αντιστοιχεία με την προσπάθεια. Υπάρχει μια μεταβλητή και διαφορετικότητα στις διάφορες GSA και μετά από την πρώτη περίοδο όπου πήγαμε ε, στα 40 χιλιοστά ή σε εκείνη τη ρομποειδή των 50 χιλιοστών φαίνεται να υπήρχε μειώση των αλλιευμάτων όσον αφορά το βάρος, αλλά μεγαλύτερη αξία όσον αφορά το μέσο μέγεθος ε, του προϊόντος, που δηλαδή έτσι πετύχαινε και καλύτερες τιμές. Αλλά μετά από μια πρώτη περίοδο αυτής της εξέλιξης, σταθεροποιήθηκαν και πάλι οι, τα αλλιεύματα τόσο όσον αφορά το βάρος ε, όσο και την τιμή όπου ήταν χαμηλότερα τελικά τα λιμάνια ε, το ευρωπαϊκό μάτι όπως αποκαλείται ε, οδήγησε σε αύξηση του μέσου μεγέθους, μείωση της παραγωγής, η αγορά πλήρωνε περισσότερο αυτά τα μεσαία μεγέθη σε μια πρώτη φάση και φαινόταν δηλαδή ότι τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα. Όμως μετά αυτά τα μεγαλύτερα μεγέθη ξαναμειώθηκαν και ξανασταθεροποιηθήκαμε σε μια τάση όπου τόσο, στην ε, τόσο η Ιταλιεύμα, τόσο και το γενικότερο βάρος μειώθηκαν. Ήταν τώρα σημαντική, σημαντικά εκεί απώλεια για τα μαλάκια και για τα κεφαλόποδα που έχουν ε, μικρό ζωτικό κύκλο και περνάνε από μεγαλύτερα μάτια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να τα ξαναπιάσει μετά όταν έχουν μεγαλώσει, απλώς χάνονται. Δηλαδή, υπάρχει ένα τμήμα αυτού του προϊόντος το οποίο χάνεται ε, οριστικώς. Και αν συγκρίνει κανείς με τον Ατλαντικό θα, πρέπει, θα διαπιστώσει ότι τα είδη της Μεσογείου έχουν διαφορετική βιολογία από ότι αυτά του Ατλαντικού. Οι κύκλοι ζωής ε, είναι διαφορετικοί όσον αφορά το χρόνο και τα χαρακτηριστικά τους. Ε, σε σχέση δηλαδή με τα ψάρια του Ατλαντικού ή της Μαύρης Θάλασσας. Δεν πρέπει δηλαδή α, να τα αναμειγνύουμε και να συγκρίνουμε αυθαίρετα. Τώρα, αυτό το ευρωπαϊκό μάτι που υποτίθεται ότι είναι πιο επιλεκτικό στην ουσία δεν αφήνει να περνάει ολόκληρο το προϊόν, αλλά να είναι χτυπημένο, γιατί το προϊόν που φτιάνει στο δίχτυ χτυπά σε ένα άλλο ψάρι που έχει ήδη πιαστεί και έπειτα ξαναβγαίνει από το δίχτυ είναι ήδη χτυπημένο, είναι προβληματικό και κάποιος βιολόγος θα είναι εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα, πάντως δεν έχει πολλές ελπίδες να επιβιώσει αυτό το είδος που έχει ήδη χτυπηθεί. Είναι πολύ εύκολο αν να το διαπιστώσει αυτό κανείς, άμα παρακολουθήσει λίγο ε, το ψάρεμα. Κάποτε οι γλάροι φτάνανε τσούρμο πάνω από τα ψαράδικα μόλις τελείωνε το ψάρεμα. Τώρα ακολουθούν τα δίχτυα γιατί αφήνουν πίσω τους ένα σωρό ψόφια ψάρια ή ε, ψάρια που είναι χτυπημένα. Επίσης, στην Αδριατική αυτή η, μη, η δυνατότητα, μάλλον το ότι δεν δόθηκε δυνατότητα εξαίρεσης, δεν επέτρεψε την ε, αλίευση μικρών ψαριών όταν είναι ενήλικα. Νομίζω πως μια αντιπροσωπεία σας επισκέφθηκε το λιμάνι της Κιόντζα πριν από λίγο καιρό και μίλησε με τους αλίες που εποχιακά ψαρεύουν ε, αυτό το είδος ε, ή ε, μοσκαρτίνη, μικρά ψαράκια δηλαδή, τα οποία είναι μικρά ακόμα και όταν είναι ενήλικα και είδαν ότι πια δεν μπορούσαν να δουλέψουν για αυτά τα είδη. γιατί είναι είδη που δεν μπορούν να ληφθούν ούτε με κάποιον άλλο εξοπλισμό. Και αυτό ήταν αρνητικό αντίκτυπο λοιπόν για τι αλληλευτικέ δραστηριότητε. Μια άλλη ομάδα αρνητικών επιπτώσεων ήταν βέβαια η αύξηση των προστήμων, ε, το, της τιμής των, της χορήγησης αδειών. Ο ελεγκτικός κανονισμός 1224 του 2008 ε, προβλέπει ότι αν έχει κανείς στο σκάφος δείγματα κάτω των επιτροπόμενων μεγεθών θεωρείται σε σοβαρή παράβαση όπως η αλληλεία άνευ αδείας. Δηλαδή ε, τι, τι ποινή πρέπει να επιβάλλεται και τι ποινή θανατική στην ουσία αφού είναι αυτό να το σκεφτούμε, γιατί η αλίευση μικρότερων ψαριών ε, από το επιτρεπόμενο ε, γίνεται ακόμα και με νόμιμα δίχτυα. Πάνε δηλαδή οι αλίες ψαρεύουν με νόμιμα δίχτυα. Αν όμως τους πιάσει ο έλεγχος με ένα ψαράκι μικρότερο, θεωρούνται μεγάλοι παραβάτες, σύμφωνα με τον 1224, τους βάζουν πρόστιμο, τους παίρνουν την άδεια και μετά, το, ή μάλλον τους βγάζουν πόντους από την άδεια και ξέρουμε ότι μόλις αφαιρεθούν κάποιοι πόντοι από την άδεια, ε, τους στερείται. Αυτά λοιπόν όλα θα πρέπει να αλλάξουν με τη μεταρρύθμιση. Διότι η υποχρέωση εκφόρτωσης ακόμα και των παραλιευμάτων σημαίνει στην ε, Μεσόγειο ακριβώς το προϊόν μικρότερο του μεγέθους που βγαίνει εκτός από άλλα ε, προϊόντα τα οποία όπου, δεν επιτρέπεται η λήψη. Αυτή τη στιγμή μόνο ο μπλε, ο, τόνος είναι αυτός που επιτρέπεται. Να. Ε, αυτός είναι το μόνο είδος που δεν επιτρέπεται να λιεύεται. Δεν, δεν, δεν, πρέπει να φτάσουμε στο παράλογο, όπου δηλαδή θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αρχίζουν να αυτοκαταγγέλλονται. τώρα δεν νομίζω ότι θα το κάνουν αυτό οι ψαράδες, θα πηγαίνουν να λένε «Να, εμείς πιάσαμε μικρότερα ψάρια». Τώρα, όταν μιλάμε για ελάχιστα μεγέθη και για μηδενική ανοχή ε, της ε, ε, των αλλιευμάτων. Ε, το άλλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα των κοχυλιών, ας πούμε, στην Αδριατική. Γίνεται συγκεκριμένη διαχείριση, γιατί εκεί υπάρχουν όμιλοι που αλλιεύουν μαζί, ε, σπέρνουν στην ουσία μαζί, γίνεται εκ περιτροπής ε, αλληλεία, αφήνουν το προϊόν να φτάσει στο εμπορικό του μέγεθος κτλ. κτλ. Πάντως είναι στόκο στο οποίο υπάρχει διαχείριση, γιατί για τα κοχύλια αυτά υπάρχει το ελάχιστο μέγεθος των 25 χιλιοστών. Αν η ακτοφυλακή βρει ένα κοχυλάκι μικρότερο, μπαίνει σε εφαρμογή αυτός ο μηχανισμός που σας θύμισα. Δηλαδή πρόστιμο, κατάσχεση του προϊόντος, πόντι ε, στην, ε, στην άδεια. Μα τι νόημα έχει να εφαρμόζονται ελάχιστα μεγέθη εκεί όπου υπάρχει διαχείριση των αποθεμάτων. Δεν θα ήταν λογικό να εφαρμόζεται στα διβάλβιδα μαλάκια αυτό που ισχύει για, το, για τα μικρά πελαγικά όπως οι ατζούγες και οι, σαρδίν, ε, οι σαρδέλες, με συγχωρείτε, όπου Δηλαδή, αντί για το ελάχιστο μέγεθος του κάθε ενός ψαριού, να υιοθετείται, για παράδειγμα, ο μέγιστος αριθμός ε, ατόμων ανά κιλό. Για τις ατζούγες δεχόμαστε τα 110 άτομα στο κιλό, για τις σαρδέλες 55 άτομα το κιλό, ενώ για τα κοχύλια δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί σε 30 σάκους που ψαρεύει ένα σκάφος το χρόνο, αν υπάρχει ένα, μία, ένα ή δύο κοχύλια 24 χιλιοστών, ενώ το επιτρεπόμενο είναι 25, του κάνουν κατάσχεση και του βάζουν και ένα πρόστιμο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια λύση προσαρμογής, γιατί ε, θα πρέπει να λογαριάσουμε με μια πραγματικότητα που έχει προχωρήσει εντωμεταξύ και δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες άλλων ελάχιστων μεγεθών που αφισβητώνται όπως ας πούμε στα Στακός ή άλλα είδη. Να... Και αυτά τα χρησιμοποιούν, ε, τα ψαρεύουν πολύ και οι Ισπανοί συνάδελφοι. Φαντάζομαι θα το αναφέρουν και εκείνοι. Και τώρα για να μιλήσουμε για τις ελάχιστες αξίες απόστασης από τις ακτές και βάθος, όπως ορίζονται από το άρθρο 13 που προβλέπει δυνατότητες εξαίρεσης. Όμως μόνο για μια σειρά συγκεκριμένων πρέπει να μάλλον πληρούνται μια ολόκληρη σειρά όρων. Θυμίζω ότι οι αποστάσεις αυτές από τις ακτές αφορούν και έχουν καθοριστεί μάλλον με βάση το βάθος. Πριν από αυτόν τον κανονισμό έλεγε ότι έπρεπε να λιεύει κανείς μόνο έξω από τα, πέρα από τα τρία μίλια και σε κάθε περίπτωση όχι μέσα στο βαθμετρικό, στη βαθμετρική ζώνη των 50 μέτρων. Αυτό σημαίνει πως εάν δεν έχω μια εξαίρεση δεν μπορώ να πλησιάσω 1,5 παρα, ε, περισσότερο από 1,5 μίλι από μια βραχώδη ακτή. Ε, ε, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ψαρέψω τίποτα. Το να, πάρει, να πετύχει κανείς όμως εξαίρεση είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορεί δηλαδή να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Μιλάμε για, ευρύ, ε, για τις ευρείες ζώνες ε, και όχι για τις ε, ζώνες όπου υπάρχουν συγκεκριμένες προεξοχές και ας λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κλειστές ε, θαλάσσιες περιοχές που είναι άλλη υπόθεση πάλι. Έχουμε λοιπόν θέμα όσον αφορά την απόσταση από τις ακτές και όσον αφορά τα σειρώμενα δίχτυα ορίστηκε η απόσταση στα 0,3 μίλια. Θυμίζω όμως ότι υπάρχουν κάποια διβάλβιδα μαλάκια τα οποία είναι εμπορικό είδος και που ζουν εντός αυτός της ζώνης. Το είδος ένσις μίνορ, εμείς ε, το λέμε σωλήνα, το οποίο δεν υπάρχει πέρα από αυτή την, έξω από αυτή τη ζώνη των 0,3 μιλίων. Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να βρούμε εξαίρεση για να μπούμε μέσα πιο, πιο κοντά στις ακτές. Λοιπόν, πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία εδώ θα ήταν ε, λογικό. Τώρα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εξοπλισμών. Είναι, αμφισβητείται αυτός ο κανονισμός από πολλές ενώσεις αλλιέων, γιατί σε σχέση με το μεγάλο πλούτο των ε, αλληλευτικών εξοπλισμών, κυρίως της, της μικρής αλίας που ήταν στην ουσία η βαθιά σοφία των αλλιέων, που προσαρμοζόταν κάθε φορά το ψάρι που έπρεπε να αλλιεύσει ακόμα και εποχιακά. Κάθε φορά προσάρμοζε τον εξοπλισμό του. Ο πλούτος λοιπόν αυτός στην ουσία ε, καταργήθηκε γιατί αυτός ο κανονισμός επέβαλε ένα είδος ε, που πιστεύοντας ότι η Μεσόγειος, όπου είναι πολύ διαφορετική η κουλτούρα της αλληλείας ανάμεσα στην, στην ακτή της Ανδαλουσίας μέχρι την Ελλάδα, περνώντας και από την Αδριατική, ότι όλα αυτά μπορούσαν να γίνονται με βάση τους ίδιους κανόνες. Και εδώ πιστεύουμε πως ε, έγινε μέγας εξαναγκασμός, γιατί υπάρχουν ε, πτυχές όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα, τις τεχνικές ιδιαιτερότητες που δεν έχουν να κάνουν ε, καθόλου με την επιλεξικτικότητα Ας πούμε, για το μέγεθος του ματιού. Εντάξει, μπορεί να σχετίζεται με την επιλεκτικότητα του εξοπλισμού. Αλλά τώρα όταν μιλάμε για παραγάδι, τι σημασία έχει άμα είναι 5 χιλιοστά ή 3 χιλιοστά. Δηλαδή σπάει συχνότερα στην ουσία. Ότι Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο κόστος διαχείρισης και περισσότερα προβλήματα για τις εταιρείες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επιλεκτικότητα, γιατί και όταν κανείς τραβά ένα σάκο πιο, ευ, ε, πιο έθραυστο, το προϊόν ε, καταστρέφεται ε, και το να βλέπετε να σπάει ένα δίχτυ δεν εφαλεί ούτε την εταιρεία ούτε τη διατήρηση του είδους. Αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες που επαναλαμβάνω, χωρίς να χρειάζεται να γίνει καμιά φοβερή και τρομερή επανάσταση, θα πρέπει να τα ξαναδούμε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Γιατί είπατε ότι πρέπει να περιμένουμε τρία χρόνια από την πλήρη έναξη ισχύω του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Μα τα τρία χρόνια, ε, για, όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία του κανονισμού, έκλεισαν τα τρία χρόνια τον Μάιο του 2013. Όσον αφορά τη διαχείριση, όχι, αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον να αποπειραθούμε μια τεχνική επανεξέταση. Μα τι να περιμένουμε. Εδώ βλέπετε τον αντίκτυπο από την αύξηση των αλλιευμάτων, τις κυρώσεις, τη δυνατότητα ε, αλλίευσης ενηλίκων μικρού μεγέθους, ε, τη μηδενική ανοχή που, δίνει, που προκαλεί προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά κάποια προϊόντα όπως ε, το, το κοχύλι, τα κυδόνια που ανέφερα πριν. Τι ελπίζει τώρα ο τομέας μας όταν αναθεωρηθεί ε, ο κανονισμός. Καμία, όπως είπα, επανάσταση, ακύρωση ή απελευθέρωση. Αυτό που ελπίζουμε είναι να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στην ουσία. Να δούμε δηλαδή τα τεχνικά μέσα συγκεκριμένα, αυτά που τελικά φάνηκε πως ήταν τα πιο ελαττωματικά που δεν μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν και που έχουν και το μικρότερο αντίκτυπο, κατά τη γνώμη μας, για τη συντήρηση, τη διατήρηση των πόρων. Δυνατότητα εξαίρεσης. Καταλαβαίνω πως για την Κομισιόν και για πολλούς η εξαίρεση είναι ε, σαν βρισιά. Δεν πρέπει κανείς ούτε να την αναφέρει αυτή τη λέξη. Όμως, είναι ένδειξη μιας ευφυούς ευελιξίας ενός ρυθμιστικού μέσου. Εκεί όπου υπάρχει αιτιολογημένη εξαίρεση, το να δοθεί εξαίρεση σημαίνει στην ουσία ότι επιβεβαιώνεται η ισχύ του μέτρου ε, με προσπάθεια να αναιρεθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου μέσου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πιστεύουμε πως το να δοθούν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα, όπου δηλαδή ε, θα έχουμε ε, χρήστες που είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν σε αυτές τις ε, διατάξεις, όπως ας πούμε η απόσταση από την, ε, την σακτές θα πρέπει να σεβαστούμε και τα βαθμετρικά στοιχεία. Ας πούμε, στα 0,3 μίλια, αν σκεφτούμε πως αυτό το μαλάκιο δεν υπάρχει πέρα από τα 0,3 μίλια, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε πως ε, θέλουμε, θα, θα πούμε ότι είναι θέμα αρχής και τα λοιπά. Μα δεν μας ενδιαφέρει μας ε, το θέμα αρχής, μας ενδιαφέρει να υπάρχουν κανόνες που να επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλματός μας με αξιοπρεπή και κερδοφόρο τρόπο χωρίς να βλάπτουμε κανένα πόρο. Η μείωση ορισμένων ελάχιστων μεγεθών ή όπως έλεγα προηγουμένως η εισαγωγή μιας εναλλακτική, ε, όπως ο αριθμός ε, ατόμων ανακυλώ για τα χαρακτηριστικά των εξοπλισμών τέλος. Μια αναθεώρηση που, που, που επανειλημμένα ζητήσαμε ακόμα και πριν να εγκριθεί ο συγκεκριμένος κανονισμός η προσαρμογή των παραρτημάτων 1 και 2 ώστε να αποφευθούν και διατυπώσεις που είναι ακατανόητες και μη εφαρμόσιμες όσον αφορά την ε, διατήρηση των πόρων. Υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιες διατυπώσεις δηλαδή, όπως ας πούμε αυτός ο σάκος με τσέπιλι μυστήριο. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι είδους δείχτη είναι αυτό και γιατί απαγορεύεται να κάνουμε κάποια πράγματα με αυτό το είδος διχτυού που δεν το έχει κανένας. Τεχνικά χαρακτηριστικά λοιπόν να και ευχόμαστε ότι αυτή τη φορά πριν να οριστούν νέα, τεχνικά χαρακτηριστικά, να υπάρξει μια φάση μεγαλύτερης τεχνικής συνεννόησης με τον κλάδο μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπονφίλιο και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τουντέλα που είναι διευθύντρια του του Διεθνούς Ταμείου για τη Φύση, για τη Μεσόγειο. Παγκόσμιος. Παγκόσμιο Ταμείο. Όχι. Thank you, Chair. Ε, καλησπέρα, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Όπως θα αναφέρω αργότερα, η εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο έχει κρίσιμη σημασία για την υποστήριξη των πόρων, των εμβίων πόρων στην Μεσόγειο. Επιτρέψτε μου να ανατρέξω στην ιστορία, έτσι όπως την βλέπουμε βεβαίω, της εφαρμογής του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Φυσικά θα εστιάσω την προσοχή μου στο μέλλον γιατί πιστεύουμε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία από τις συγκεκριμένες συνθήκες για να εξασφαλίσουμε αηφορική αλληλεία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νέας αλληλευτικής πολιτικής. Ξεκινώ λοιπόν Όπως ε, προείπα, για μας ο κανονισμός για τη Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικό νομοθετικό κείμενο. Εμείς λάβαμε ενεργά μέρος στην τελευταία αναθεώρηση της ελευθερικής πολιτικής το 2001-2002. Υποστηρίξαμε την τροποποίηση του τότε κανονισμού για την Μεσόγειο Γνωρίζετε φαντάζομαι και τον παλιό κανονισμό που ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανεπαρκής για την διαχείριση των πόρων στη Μεσόγειο. Αποτελούσε ένα απλό άθροισμα τεχνικών μέτρων. Ήταν μια βασική θα νομοθεσία. Ήταν αδρήτη ανάγκη λοιπόν η βελτίωσή του. Όταν η Κομισιόν κατέθεσε την πρόταση κανονισμού το WWF εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί το νέο κείμενο είναι πληρέστερο μάλιστα προβλέπει και καινοτόμα μέτρα διατήρησης προστατευόμενα ενδιαιτήματα παιδεία ποσειδονίας καθώς και ασβεστολιθικά πολύματα αφικών και ούτω καθεξής εισάγει βεβαίω των θέσμα των προστατευμένων περιοχών, κάτι το οποίο ήταν καινοτόμο την εποχή εκείνη, υπό την έννοια ότι προέβλεπε τη δημιουργία διαχείρισης αναπεριοχή με βάση την βλάβη που θα μπορούσε να προκαλέσουν οι ελληνικές πρακτικές στη συγκεκριμένη όμως περιοχή. Κάτι το οποίο δεν ήταν η τρέχουσα πρακτική την εποχή εκείνη. Αυτά ήταν τα καλά Ταυτόχρονα, κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου για κάτι το οποίο θα παραλάβω αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της της εισηγησής μου. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν τα σχέδια διαχείρισης. Αυτό είναι και το κλειδί της υπόθεσης και αυτό θα μας βοηθήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων για να αντιμετωπίσουμε την υπεραλίευση στη Μεσόγειο. ποιες είναι οι αδυναμίες των σχεδίων διαχείρισης. Όλα τα σχέδια απολάβουν εξαιρέσεων και παρεκκλήσεων. Για εμάς τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εφορικής ελίας στην Μεσόγειο και εμπόδιο στην πυραλίευση. Παράδειγμα, για να θυμίσω λίγο και το ιστορικό της υπόθεσης. Εδώ διαβάζουμε κάτι το οποίο έχει ήδη ηλικία 10 ετών. Ήταν ένα από τα πρώτα κείμενα που καταθέσαμε σχολιάζοντας την πρώτη πρόταση της Κομισιόν. Ήταν Οκτώβριο του 2003 συγκεκριμένα το WWF με ανησυχία. Έλαβε το κείμενο οι επιλεκτικές παρεκκλήσεις επί διαφορών διατάξεων για τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο των μέτρων των σχεδίων διαχείρισης. Κρούμε το κοντά του κινδύνου διότι οι εξαιρέσει την να γίνουν ο κανόνας. Και παραπέμπουμε μετά στο άρθρο 17, το οποίο γίνεται μετά 19. Φαίνεται ότι μερικά σχέδια διαχείρισης έχουν καταστρωθεί με ακριβώς αυτό ως στόχο. Την εξασφάλιση δηλαδή εκτελών παρεκκλήσεων εν ώψη της έγκρισης του κανονισμού. Να είμαστε όμως δικαίοι. Δεν ήρθα εδώ για να γκρινιάξω. Είναι πολύ εύκολο να γκρινιάζει κανείς για το ένα ή το άλλο. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε με τρόπο επικοδομητικό, κατανοώντας το πλαίσιο στο οποίο επιχειρούμε. Ο κανονισμός για τη Μεσόγειο ήταν η τελευταία νομοθεσία από την εποχή του 2001-2003 και ήταν κληρονομιά της παλιάς προσέγγισης, της μικροδιαχείρισης αυτό το οποίο προσπαθούμε ακόμη να ξεπεράσουμε. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι η κεντρική μικροδιαχείριση από τις Βρυξέλλες Οικονομεύει ακριβώς την ευλογή εξορθολογισμένη διαχείριση βάσει των τοπικών συνθήκων. Οι εξαιρέσεις λοιπόν μέσω τεχνικών μέτρων στα σχέδια διαχείριση υποτίθεται ότι ένα καλό πράγμα για να εξορθολογιστεί και να είναι λειτουργικό το καθεστώ. Αυτό ήταν η λογική. Όμω, με αυτόν τον τρόπο τα σχέδια διαχείριση αντί να εστιάζονται στην αηφορική πτυχή τη αλίας αντί να προσανατολίζεται στην διατήρηση και προστασία, ζούσαν με εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων. Και αυτό είναι ακριβώς η βασική μας κριτική. Πριν από τρία χρόνια, τον Μάιο του 2010, υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δική μας αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου κανονισμού. Ε, να μην τα ξαναπώ, τα έχουμε γράψει όλα και έχει πει η Κομισιόν αυτά που είχε να πει απόψε. Πάντως ε, προέβημε σε μια επισκόπηση βάσει ερευνών που κάνουμε κατά πάγιο τρόπο σε διάφορα κράτη-μέλη. Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα κλπ διαπιστώσαμε σημαντικές παραλήψεις και αστοχίες στην προστασία των ενδιατημάτων. Έχουμε ένα σχετικό πρόγραμμα που τρέχει για όλα αυτά και ε, οι οποίε ε, αστοχίες αφορούν τις προστατευμένε περιοχές. Διαπιστώσαμε επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν καν σχέδια διαχείριση, παρά το ότι τα σχέδια αυτά ήταν υποχρεωτικά για μία τριετία. Επίσης, διαπιστώσαμε παρατυπίες στην εφαρμογή. Και για να είμαι ποιηκής ε, αυτό οφείλεται, για να το πω αλλιώ ε, στην έλλειψη πολιτικής βουλής από ψηλά. Μετά η διαδικασία έγκρισης των σχεδίων και το ποιος κάνει τι δεν είναι το σαφής. διπιστώσαμε λοιπόν και την έλλειψη σαφήνειας κάτι το οποίο αποτελεί και ένα από τα αίτια της αποτυχίας στον τομέα. Συμβουλεύσαμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει και κατευθυντηρείς γραμμές για την υλοποίηση της κατάστροφης αυτών των σχεδίων διαχείρισης. Επιτρέψτε μου να διαβάσω αυτήν την ε, παράγραφο, γιατί πιστεύω συμπυκνώνει με σαφέστατο τρόπο τη θέση μας. Τότε και σήμερα. Επιτρέψτε μου λοιπόν, διαβάζω. Είναι κάτι το οποίο συνταχθεί πριν από τρία χρόνια, το 2010. Εφτά ολόκληρα χρόνια μετά από το κείμενο που παρουσίασα πιο νωρίς. Πιστεύουμε ότι τα σχέδια διαχείριση πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίο λίθο τη διαχείριση τη Ελία στη Μεσόγειο. Τα ισχυρά του όμω δεν πρέπει να περιοριστούν στον παρόντο κανονισμό. Τα σχέδια δεν πρέπει να αποτελούν οδό διαφυγής από τα πρότυπα και να αποτελούν δικαιολογία ή πρόσχημα για παρεκκλήσεις. Ίσα ίσα, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, πρέπει να θέτει τα κοινά πρότυπα τα οποία θα ισχύουν για τα σχέδια και βεβαίως να εγκρίνονται τα μέτρα διαχείρισης προσαρμοσμένες στις κρατόπους συνθήκες. Τα σχέδια πρέπει να είναι υποχρεωτικά για κάθε περιοχή της Μεσογείου. Η δε επιτυχής εφαρμογή τους πρέπει να την χάνει εγγύησης από τους συγγραφείς του σχεδίου. Για αυτούς που εν τέλει το εγκρίνουν. Και εδώ αναφέρομαι και στην συνδιαχείριση. Η συνδιαχείριση είναι κλειδί για την επιτυχία της εφαρμογής κάθε σχεδίου διαχείρισης. Αυτά λοιπόν όλα τα σχέδια πρέπει να ελέγχονται, να παρακολουθούνται και να αναθεωρούνται από επιτροπές συνδιαχείρισης σε αποτελούμενες από τους εμπλεκομένους. Λοιπόν, αυτό το κείμενο συμπυκνώνει ακριβώ και το που βρισκόμαστε σήμερα. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, με βάση πληροφορίες που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώθηκε σημαντική πρόοδο στον, στο πλήθος των σχεδίων διαχείρισης και στο πλήθος των προστατευμένων περιοχών που δημιούργησαν τα κρατημέλη. Παρ' όλα αυτά, με βάση τις πληροφορίες μας, τα εγκεκριμένα σχέδια δεν εστιάζουν σε ολοκληρωμένα μέτρα για την εφορική διαχείριση των θαλασσίων πόρων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Σε ορισμένε ακραίες περιπτώσεις, και θέλω να αναφέρω ονόματα ή χώρες, απλώς επαναλαμβάνονται με τρόπο σπασμωδικό τεχνικά μέτρα, αντί για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αναβίωση, την ασύσταση των θαλασσίων πόρων, των αληφτικών πόρων. Και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που θα πρέπει να γίνει για τους ελευτικούς πόρους που έχουμε πλήξει όπως ακούσαμε και από τους αδέλφους του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Και πάλι επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα σχέδια διαχείριση. Αυτό είναι το εργαλείο το οποίο ήδη έχουμε, αλλά πρέπει να το βελτιώσουμε. Πρέπει να το ξυπήσουμε με πιο ικανοποιητικό τρόπο. Επίσης, πιστεύουμε ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα προστασία των προστατευμένων ενδιατημάτων είναι ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο της κοινή προσπάθεια το είπαμε και προηγουμένως. Ποια είναι τα θετικά λοιπόν και ποιε είναι οι προοπτικέ για το μέλλον. Ο τίτλος εδώ νομίζω τα λέει όλα. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Έτσι τελειώνει η φράση. Ο κανονισμός λοιπόν δίνει δυνατότητες για αποτελεσματική δράση, μόνον όμω και με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά θα συνοδευτούν με παρκή πολιτική βούληση στα κρατημέλη. Ακούσαμε και το παράδειγμα από την Κομισιόν λίγο πριν. Τώρα στην Καταλωνία υπάρχουν πολλές επιτροπές συνδιαχείρισης, ελίας, στην οποία συμμετέχουν ε, η διοίκηση, η ΜΚΟ, αλής, η μηχανία, κρατικές αρχές κλπ. Αυτό το σχήμα είναι ένα κοινοτόμο σχήμα και είναι εξαιρετικά επιτυχημένο. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο προέκυψε βάσει του κανονισμού. Δηλαδή τα εργαλεία υπάρχουν. Υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση και η πολιτική βούληση και έτσι το αρχικό σχήμα εξελίχθηκε σε κάτι πραγματικά καινοτόμο το οποίο εργάζεται υπέρ της αηφορικής αλίας και της προστασίας των αλιευμάτων. Και αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα της παρουσίασής μου ότι τα σχέδια διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν από εδώ και πέρα έναν ικανό μηχανισμό υλοποίησης της νέας προσέγγισης με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων και την διατήρηση των αποθεμάτων πάνω από το ελάχιστα βιώσιμα αποθέματα. Το εργαλείο αυτό, επαναλαμβάνω, υπάρχει, δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως, δεν έχει πάρει σάρκα και ωστά, αλλά θα είναι σχετικά εύκολο το εργαλείο αυτό να αξιοποιηθεί με βάση της διατάξεις και με την αύξηση των αποθεμάτων πάνω από τα ελάχιστα βιώσιμα αποθέματα. για τα επόμενα χρόνια. Όπως γράφουμε και εδώ, τα σχέδια διαχείρισης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την υλοποίηση της νέας πολιτικής. Για την μείωση, για παράδειγμα, των απορρίψεων με αυξημένη επιλεκτικότητα, καλύτερη επιλογή ελευτικών εργαλείων κλπ. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια απέτηση για όλα τα σχέδια, αλλά και για κάθε σχέδιο το οποίο θα εγκριθεί από εδώ και πέρα. Το ίδιο ισχύει και για την περιφερειοποίηση, τη λεγόμενη περιφερειοποίηση, κρίσιμο στοιχείο για την υλοποίηση της νέας ελευθερικής πολιτικής στη Μεσόγειο. Μάλιστα θα έλεγα ότι ότι τα σχέδια διαχείρισης υπό τον νέο κανονισμό ενδεχομένως αποτελούν και τη βέλτιστη ευκαιρία για την υλοποίηση εκβάθρων του νέου κανονισμού στο πλαίσιο της νέας αλληλευτικής πολιτικής. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο δρόμος. Για εμάς είναι απολύτως σαφές. Φυσικά τα εθνικά σχέδια διαχείρισης υπάρχουν και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται στο πλαίσιο του κανονισμού αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω επιτροπών συνδιαχείρισης. Και έτσι θα είναι και επιλέξιμα για ενισχύσεις από το αρμόδιο ταμείο. Κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί, θα οριστικοποιηθεί και στο πλαίσιο του επικειμένου τριμέρου τριμερούς διαλόγου. Η περιφερειοποίηση αυτή πρέπει να γίνει με την συμμετοχή του Περιφερειακού Συμβουλευτικού Οργάνου για τη Μεσόγειο και Επιτρέψτε μου να κλείσω σε αυτό το σημείο γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ήθελα να θυμίσω τα βασικά στοιχεία και μάλιστα σε έναν τόνο αισιόδοξο. Ακόμα ένα σωρό άσχημα νέα σχετικά με το που πηγαίνει η Ελία στην Μεσόγειο. Ακούμε άσχημα νέα ε, σχετικά με, το, με την κακοδιαχείριση ως τώρα, κάτι το οποίο ήταν αλήθεια σήμερα. Δεν υπάρχει καμία εμφολία περί αυτού. Όμως ας κοιτάξουμε στο μέλλον και ας δούμε τι δυνατότητες έχουμε μπροστά μας. Μάλιστα θα δείτε ότι όσο αφορά τις μελλοντικέ μας προοπτικές δεν τα έχουμε πάει και δεν τα πηγαίνουμε τόσο άσχημα. Ας κάνουμε ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε την εικόνα με το δικό μας ρόλο και ας εφαρμόσουμε τον κανονισμό με τρόπο που συνάδει με τη νέα ληφτική πολιτική. Και έτσι πιστεύω ότι θα πετύχουμε καθαρή βελτίωση και αύξηση των αποθεμάτων στην περιοχή μας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τουδέλα. Και τώρα τελευταίος προσκεκλημένος μας είναι ο Δον Χωσέ Μαρία Γκαλιάρ, πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων της Αλίας, της Αλμερίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι αντιπρόεδρος της ε, Ένωσης Αλλιέων αυτής στην ε, Αλμέρια και είναι πολύ σημαντικό για μας ε, να έχουμε τη δυνατότητα να σας μιλήσουμε εδώ σήμερα και να σας δώσουμε τη δική μας εικόνα της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο Ισπανικός αλλιευτικός στόλος στη Μεσόγειο. Μπορούμε να σας αναφέρουμε τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Θα σας πούμε επίσης τι κάνουμε για να πετύχουμε βιώσιμη αλληλεία, κοινωνική ανάπτυξη, να διασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Θέλουμε να έχουμε βιώσιμη αλληλεία και να το πετύχουμε αυτό με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι συμβατά. Με κάποιες από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Κομισιόν. Παρακολουθούμε τα όσα λένε τα διάφορα θεσμικά όργανα και θέλουμε να έχουμε μια αλληλευτική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του τομέα μας. Θέλουμε επίσης να έχουμε κανόνες τους οποίους να μπορούμε να ακολουθήσουμε. Να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το τον Ισπανικό στόλο και είναι στοιχεία του Νοεμβρίου που θα σας δώσουν μια εικόνα της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.762 σκάφη, 58.454,59 ε, τόνοι και 236.648 κιλοβατόρες. Τα περισσότερα σκάφη αυτά είναι τράτες αλλά θα πρέπει να σας παρουσιάσουμε και την εξέλιξη από το 2006 και μετά, από τότε που υιοθετήθηκε ο κανονισμός για τη Μεσόγειο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν γίνει διάφορες αλλαγές για να προσαρμοστούμε στους πιο αυστηρούς κανόνες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο της αλλιευτικής προσπάθειας. Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Στον επόμενο πίνακα λοιπόν βλέπετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στον στόλο μας. Από το 2006 και μετά είχαμε 3.098 σκάφη τότε. Και με επιδοτήσεις έχουμε μειωθεί τώρα στα 2.762 σκάφη, μία πτώση της τάξης του 30% στον αριθμό των σκαφών. Και αναφέρομαι στο σύνολο των ειδών των σκαφών. Από την Ανταλουσία, τη δική μου περιφέρεια βλέπετε ότι είχαμε μείωση και σε αυτήν την αυτόνομη περιφέρεια. Έχουμε μείωση της τάξης του 40%. 2% στις στράτες. Και επίσης, όπως αναφέρθηκε πριν, πιστεύουμε ότι βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον η τάση θα είναι να μειωθούν περισσότερο τα σκάφη του αλλιευτικού στόλου. Επίσης, να αναφερθώ τώρα στην εφαρμογή του κανονισμού 7 χρόνια μετά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει αναθεώρηση και να εξεταστούν ποιες ήταν οι επιπτώσεις για τον τομέα μας. Κάθε κανονισμός πιστεύω πρέπει να αναθεωρείται και να βελτιώνεται. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να γίνει και με τον κανονισμό για τη Μεσόγειο. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν διάφορα στοιχεία και διάφορα είδη εξοπλισμού. Όσον αφορά λοιπόν τις στράτες, αυτή ήταν η πιο σκληρή προσαρμογή που έπρεπε να κάνουμε και ο κύριος Μπορφίλιο αναφέρθηκε σε αυτό. Έγιναν λοιπόν τροποποίησεις όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος του ματιού, καθώς και το πάχος του νήματος. Όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος ματιού για τα δίχτυα τράτας, και ιδιαίτερα για τα σειρώμενα δίκτυα, στο άρθρο 14 προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι την 31η Μαΐου του 2010. Μετά από αυτό θα έπρεπε να ε, αντικατασταθούν τα δίχτυα από δίχτυα με τετράγωνο μάτι μεγέθους 40 χιλιοστών. Έχουμε τον κανονισμό 1343 του 2011 που έχει επιφέρει περαιτέρω αλλαγές και το άρθρο που μας ενδιαφέρει κυρίως εδώ έχει αποτελήσει αντικείμενο διαφόρων ερμηνεών. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες σε σχετικά με το μέγεθος ματιού στο άρθρο αυτό. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο για μας να εφαρμόσουμε τις αλλαγές αυτός, ε, τις αλλαγές αυτές, καθώς και να επιβεβαιώσουμε το μέγεθος του ματιού των δικτύων που χρησιμοποιούνται, διότι όπως σας είπα υπάρχουν διάφορες ερμηνείες του κανονισμού αυτού. Για τους λόγους αυτούς υπήρχε ανασφάλεια στον τομέα της αλληλείας σχετικά με το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν για να γίνει η προσαρμογή στο νέο κανονισμό. Σε διάφορες περιστάσεις λοιπόν έπρεπε να αλλάξουμε εξοπλισμό. Ανάμεσα στο 2010 και το 2013 λοιπόν, δύο φορές έγιναν αλλαγές στους σάκους λόγω των διαφόρων ερμηνεών του κανονισμού. Έχουμε πληρώσει όμως τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την νομοθεσία αυτή. Νιώθουμε όμως ότι θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα εάν ήταν πιο σαφής η διατύπωση των διαφόρων κανόνων που συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό αυτών. Όσον αφορά το πάχος του νήματος, αυτή είναι μια από τις βασικές ανησυχίες μας. Υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί λόγοι γιατί αποτελεί πρόβλημα αυτό. και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να συμμορφωθούμε με τους κανόνες, αλλά η πρακτική αυτή είναι δύσκολο θέμα για τις αλληλευτικές δραστηριότητες και των εθνικών φορέων μας και στο ΡΑΚ της Μεσογείου έχουμε παρουσιάσει τις θέσεις μας για το συγκεκριμένο σημείο. Μας έχουν ζητήσει στοιχεία γιατί αυτό αποτελεί πρόβλημα για μας. Και αυτή τη στιγμή εκπονείται μελέτη η οποία θα διαρκέσει πολύ χρόνο και στοιχίζει και πολύ. Η οποία όμως θα δείξει μια και καλή τα επιχειρήματα στα οποία εμένουμε. Λέμε λοιπόν ότι το βάρος και η ανθεκτικότητα του νήματος δημιουργούν προβλήματα. Κάτι που έχει και οικονομικό αντίκτυπο και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες αυτοί όσον αφορά τα 6 χιλιοστά για το πάχος του νήματος. Θα σας παρουσιάσουμε τεχνικά στοιχεία να σας το αποδείξουμε αυτό. Και Επίσης, ε, όσον αφορά την ε, απόσταση από την ακτή και το βάθος. Γενικά η σε όλο τον κανονισμό είναι δύσκολο να εφαρμοστούν οι σχετικοί κανόνες και είναι θέμα και γεωγραφικό που έχει να κάνει με τις διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι πιο χρήσιμο να μιλάμε για βάθος παρά για απόσταση από την ακτή. Αυτού του τύπου εξοπλισμός είναι από τους καλύτερους όσον αφορά τη ζημιά που κάνει στη θάλασσα. Θέλουμε να προστατεύσουμε το βυθό και δεν καταλαβαίνουμε το θέμα της απόστασης. Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη τις διάφορες περιοχές και τα διάφορα είδη ακτών, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά παντού. Είναι δύσκολο θέμα λοιπόν η απόσταση Και όσον αφορά την απόσταση από την ακτή, το θέμα είναι βέβαια ότι δεν θέλουμε να αλλιεύουμε νέους θαλάσσιους οργανισμούς, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος των ψαριών που αλλιεύονται στις περιοχές αυτές. Σε όλες τις διάφορες συναντήσεις λοιπόν που είχαμε με την Κομισιόν, εξετάζουμε το μέγεθος δύο συγκεκριμένων ειδών του σαφριδιού και της Τσιπούρας. Και δεν ξέρουμε πώς αποφασίστηκε το συγκεκριμένο μέγεθος για τα ίδια αυτά στην Ισπανία. Γύρω από το Γιβραλτάρ έχουμε σχέδιο αποκατάστασης για τα δύο αυτά είδη και τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και γι' αυτό είναι πολύ περίεργο το ότι το ελάχιστο μέγεθος που έχουμε στον κανονισμό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο σχέδιο αποκατάσταση. Παρακαλούμε την Κομισιόν λοιπόν να ανεθεωρήσει αυτά τα ελάχιστα μεγέθη. Όσον αφορά τα παραγάδια επιφανεια, εφαρμόζουμε όλους τους κανόνες της ICAT, αλλά είναι δύσκολη η εφαρμογή όσον αφορά τον ξηφία και τον ερυθρό τόνο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα έχει πει η Επίτροπος. Παρά τις επιστημονικές συμβουλές δεν είδαμε καμία αύξηση της ποσόστοσης του ερυθρού τόνου, παρότι έχει υπάρξει αποκατάσταση. Εμείς στον τομέα της αλληλείας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ανάλογα με την κατάσταση των αποθεμάτων αλλά ζητούμε, απαιτούμε όταν εκπονούνται αυτές οι εκθέσεις, σας παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη σας τις πληροφορίες που έχουμε εμείς στα χέρια μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο στόλος παραγαδιάρικων στην Μεσόγειο έχει εφαρμόσει κάποιες αλλαγές ανάλογα με τους κανόνες της ICAT και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχει γίνει προσπάθεια για να προστατευτούν οι νέοι θαλάσσιοι οργανισμοί. Ο Ισπανικός στόλος έχει ακολουθήσει λοιπόν τις συμβουλές αυτές και τα τελευταία χρόνια φροντίσουμε να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην αλλιεύουμε νέους θαλάσσιους οργανισμούς και σχετικό Ινστιτούτο στην Ισπανία ασχολείται με το θέμα. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε περισσότερους ε, νέους αλλιώς οργανισμούς. Ε, υπάρχουν δηλαδή βιολογικοί λόγοι για τις αλλαγές αυτές. Και επίσης στο άρθρο 19 λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης ανάλογα με τα διάφορα είδη αλληλείας η Ισπανία σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Έχει δημοσιεύσει σχέδια διαχείρισης αλληλείας για το σύνολο των περιοχών της Ισπανίας, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την Μεσόγειο. Το 2006, πριν υιοθετηθεί ο οργανισμός αυτός από την Κομισιόν, είχαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης για την Μεσόγειο, που συμπεριελάμβανε αυτά τα πεδία αναπαραγωγής και είχαμε και επίσης περίοδο πάυσης της αλληλείας. Στα επόμενα χρόνια εκπονήσαμε διάφορα σχέδια διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό και το τελευταίο δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 για τα γρηγρή, την τράτα και ε, σταθερό εξοπλισμό περιορισμένου μεγέθους. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτό που παρουσίασε η Κομισιόν για την Μεσόγειο, συγκεκριμένα για την περιοχή της Ανταλουσίας. Στον χάρτη που μας δείξατε, δεν είδα το σκούρο μπλε χρώμα που θα έπρεπε να υπάρχει στην περιοχή αυτή. Φαινόταν σαν να υπάρχει τέτοιο σχέδιο σε άλλα μέρη της Μεσογείου, όμως, όμως όχι γύρω από την Ανταλουσία. Αυτό μάλλον θα ήταν λάθος κατά την κατάρτιση των διαφανειών. Ο τομέας αλίας λοιπόν της Ισπανίας συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και τους κανόνες της ΣΤΕΚΦ και έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά από τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς και από τους επιστήμονες και από εμά επίσης. Το Ισπανικό Ινστιτούτο Οκεανογραφίας έχει δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα πιο ευάλωτα αλλά και πιο πολύτιμα εμπορικά είδη. Και στόχος ήταν να εξεταστούν τα βιολογικά δεδομένα για τη διάρκεια εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης. Εξετάσαμε λοιπόν το θέμα της νησιμότητας αλλά και άλλους παράγοντες. Εξετάσαμε το θέμα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Και επίσης εξετάσαμε και τι έχει γίνει από διάφορες ομάδες εργασίας από το 2010 και μετά. Εξετάσαμε λοιπόν τα περιοριστικά μέτρα και σύμφωνα με το σχέδιο αυτό Έχουμε εκπονήσει και ένα σχέδιο παρακολούθησης και συνέχειας. για να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τους πόρους, ώστε να μπορέσουμε, εάν είναι απαραίτητο, να υιοθετήσουμε μέτρα, ώστε ανα πάσα στιγμή να μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές. Όσον αφορά τη νέα κοινή αλλιευτική πολιτική στο ισπανικό κομμάτι της Μεσογείου η αλληλεία είναι ένας από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες Έχουμε εξετάσει λοιπόν τα διάφορα σημεία της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, προσαρμογή του στόλου τρίτες χώρες, προστασία των χώρων αναπαραγωγής. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να γίνει η απλοποίηση και ενοποίηση ώστε να έχουμε βιώσιμη αλληλεία. Η παραδοσιακή παράκτη αλληλεία είναι πολύ σημαντική στην περιοχή μου. Θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό και να την στηρίξουμε περισσότερο στη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική. Στη νέα λοιπόν ε, κοινή αλληλευτική πολιτική και στο νέο πλαίσιο, το οποίο θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια, δεν υπάρχουν μέτρα βελτίωσης ε, της ζωής των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλληλεία. Ο τομέας μας είναι στρατηγικός ε, κοινωνικά και οικονομικά. και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει βιωσιμότητα, αηφορία. Πιστεύουμε όμως επίσης ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν λαμβάνονται υπόψη στη νέα κοινή αλλιευτική πολιτική. Υπάρχει η περιβαλλοντική σταθερότητα, η οποία φυσικά είναι πολύ σημαντική, η οικονομική και κοινωνική ε, σταθερότητα όμως δεν φαίνονται να θεωρούνται εξίσου σημαντικές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε τους αλληλευτικούς πόρους στο μέλλον, ώστε να έχουμε βιώσιμη και κερδοφόρα αλληλεία και να προστατεύσουμε το περιβάλλον ταυτόχρονα. Στον βασικό κανονισμό δεν γίνεται αναφορά των παραδοσιακών της παραδοσιακής παράκτειας αλληλείας. Και γίνεται διάκριση ανάμεσα με το μήκος του σκάφους, αλλά αυτή είναι η μόνη διάκριση που γίνεται. Θεωρούμε ότι αν γίνεται τέτοιου τύπου διάκριση θα πρέπει να παρέχεται και οικονομική και κοινωνική υποστήριξη. Επίσης, η κατηγοριοποίηση του στόλου ανάλογα με το μήκος του σκάφους που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη μα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μα. Απλά θα ήθελα να πω ότι η διάκριση που κάνει η Κομισιόν στα σκάφη άνω και κάτω των 12 μέτρων σημαίνει ότι έχουμε 650 σκάφη τα οποία δεν ταιριάζουν στα μέτρα αυτά και θεωρούμε ότι το μήκος του σκάφους δεν αρκεί για να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στη βιομηχανική και την παραδοσιακή αλία. Υπάρχουν επίσης παράγοντες όπως είναι το πόσο φρέσκο είναι το ψάρι και η αλληλεία της ημέρας Υπάρχουν πολλέ οικογένειε που ασχολούνται με την ε, παραδοσιακή αλληλεία. Η ισπανική παράκτια παραδοσιακή αλληλεία είναι σημαντικό τομέα και παρέχει ένα βιώσιμο μοντέλο για την αλληλεία και αποτελεί μέρο τη κοινωνική και παραδοσιακή και πολιτιστική υφή των αλληλευτικών κοινοτήτων. Αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί η Κομισιόν δεν υιοθέτησε το μέτρο διάκρισης, ως μέτρο διάκρισης στα 15 ή 16 μέτρα μήκους. Ε, γιατί κάνετε τη διάκριση στα 12 μέτρα. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στα σκάφη και ανάμεσα στους λιμένες. Μας απασχολούν πολύ οι επιστημονικές σύμβουλες για το θέμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για τα διάφορα είδη και τα διάφορα αλλιευτικά πεδία. Θα ήθελα να τονίσω τον σημαντικό ρόλο του Ισπανικού Ινστιτούτου Οκεανογραφίας λόγω των δεδομένων για τα βαθύβια και βελτοπελαγικά είδη. Σε τακτική βάση πραγματοποιούνται μελέτες για τα πιο σημαντικά είδη, όπως είναι οι σαρδέλες, τον μερλούκιο και άλλα είδη και πρέπει να έχουμε πάντα επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία. Η επιστημονική κοινότητα έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη του τομέα και ο τομέας αυτός να αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες κομμάτι της οικονομίας. Όσον αφορά τις απορρίψεις, Υπάρχει το θέμα των κλειστών περιοχών, των ποσοστώσεων και του μεγέθους των ηχθείων. Απορρίψεις όμως μπορεί να πραγματοποιούνται και επειδή δεν μπορούν να απολυθούν τα ψάρια. Οι απορρίψεις όμως αποτελούν σπατάλη πόρου, σημαντικού πόρου και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαχείριση. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι κάτι που αφορά το σύνολο του στόλου που αλλιεύει στη Μεσόγειο. Δεν ξέρουμε τι, πώς θα πρέπει να τροποποιήσουμε τα σκάφη ώστε να μπορούν ε, να κρατάνε όλα τα ψάρια που αλλιεύονται. Η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη της στα διάφορα είδη του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Στην Ανταλουσία μπορεί να έχουμε 100 είδη, τα 50 από αυτά να είναι εμπορικά. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε τέλος απορρίψεις, ε, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό βαθμιαία και μακρυπρόθεσμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε είδος προς είδος και να δούμε τι συνέπειες θα υπάρξουν και θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλες τις απαραίτητες επιστημονικές πληροφορίες για να αποφύγουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Φυσικά πρέπει να διατηρήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον γενικά, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πολιτικές ώστε να διασφαλίσουμε την αποκατάσταση των αλλιευτικών αποθεμάτων και των ζωνών αναπαραγωγής. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με τρόπο βιώσιμο. Συμφωνούμε με, όλα, με όλους αυτούς τους στόχους και πιστεύω ότι η Ισπανία δίνει καλό παράδειγμα. Φροντίζουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε, φροντίζουμε η αλία μας να είναι απολύτως συμβατή με τα μέτρα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη διατήρηση της αλληλείας. Και για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή του τομέα στην επιστημονική εκτίμηση των πόρων. Μας περιμένουν ε, σημαντικές προκλήσεις, μεγαλύτερες από ποτέ. Θέλουμε λοιπόν να φροντίσουμε να μπορούμε να διατηρήσουμε τον αλλιευτικό μας στόλο. Είναι όμως κάτι το οποίο δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Ο στόλος με τράτες στη Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουν μήκος 15 με 24 μέτρα, αλλιεύουν καθημερινά. Συνήθως ε, απουσιάζουν από τους λιμένες επί 12 ώρες. Γιατί πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι τόσο σημαντική η αλία μετράτες; Κανένα είδος εξοπλισμού δεν φταίει, φταίει η χρήση που γίνεται του εξοπλισμό αυτού. Μπορεί λοιπόν να είναι περισσότερο ή λιγότερο βλαβερό κάποιο είδος εξοπλισμού. Εάν υπάρχουν ε, λοιπόν ευαίσθητα ε, οικοσυστήματα όπως είναι τα σφουγγάρια, τα κοράλια κλπ. θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Οι τράτες μας χρησιμοποιούνται σε αμμόδι βυθό όπου δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο. Είναι κάτι που ρυθμίζεται από διάφορους φορείς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την GFCM και άλλους φορείς. χρησιμοποιούμε μέθοδο που μας επιτρέπει να αλλιεύσουμε ε, οικονομικά και κοινωνικά σημαντικά είδη και αποτελεί πηγή θέσεων απασχόλησης άμεσα και έμεσα οι αλία μετράτες. Επίσης μας παρέχει προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ε, μεσογειακής δίαιτας, της μεσογειακής διατροφής. Και κλείνοντας ε, να πω για την αναθεώρηση του κανονισμού ότι θα θέλαμε το μέγεθος ματιού 15 χιλιοστών που ε, θα θέλαμε να δούμε, ελάχιστο μέγεθος ματιού 15 χιλιοστά, ε, θα θέλαμε να δούμε μέτρα όσον αφορά το σαφρίδι, τον ορισμό της παραδοσιακής παράκτεια αλληλείας που να ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα ε, στον τομέα, Καλύτερε επιστημονικέ συμβουλέ ε, καθώ ε, και γενικότερα ενίσχυση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Αφού ακούσαμε όλους μας τους προσκεκλημένους, να ανοίξουμε ένα γύρο παρεμβάσεων, όπως ήθιστε. Ε, ποιοι βουλευτές θέλετε να πάρετε το λόγο. Κυρία Φράγα, σας ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Τουδέλα και είναι η εξής. Ποιος είναι ο αρνητικός αντίκτυπος της πολιτικής απορρίψεων ε, στην Μεσόγειο όσον αφορά την πολιτική ε, διατήρησης και αυτή η πολιτική μπορεί να έχει επιρροή στο θέμα των απορρίψεων όπως ορισμένοι ρωτήσαμε. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η γνώμη σας. Κυρία Λόβιν, ας κάνουμε το εξή. σα, ακούσουμε όλε τι ερωτήσει και στο τέλος θα απαντήσετε όλοι. Κυρία Λόβιν, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Τουδέλα. Η οργάνωσή σας μίλησε για τον κίνδυνο της μικροδιαχείρισης, micromanagement, με τον κοινό κανονισμό για τη Μεσόγειο. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το πώς ε, τα πάει ο κανονισμός. Ακούσαμε από το Σαλής ότι διαμαρτύρονται πολύ, ότι είναι εξαιρετικά λεπτομερείς οι κανόνες. Εσείς πιστεύετε πως αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί μέσω επιτροπών συνδιαχείρισης εντελώς. Πιστεύω πως η ιδέα αυτή είναι πολύ ελκυστική, επιτροπές συνδιαχείρισης ή κάποιες μορφές αυτών. Είδαμε ένα σύστημα παρόμοιο στις ΕΠΑ, όπου φαίνεται να λειτουργεί, γιατί δεν είμαι και εμπειρογνώπνα στο θέμα, αλλά έχω την εντύπωση πως λειτουργεί ε, εκεί αυτό το σύστημα. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τους άλλους ομιλητές, τον κύριο Μπομφίλιο και τον κύριο Γκαλάρτ από την Ισπανία. Ποιες είναι οι δικές σας απόψεις για τις επιτροπές συνδιαχείρισης. Εσείς θα ήσασταν έτοιμοι να κάνετε μια προσπάθεια και να δημιουργήσετε τέτοιο είδος ε, πρωτοβουλίες. Στη Μεσόγειο και στον κύριο Μπομφίλιο θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω γιατί θέσατε ένα πολύ καλή ερώτημα στην αρχή της παρέμβασής σας. Είπατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι προφανές πως κάτι δεν πάει καλά. Αλλά τι δεν πάει καλά. Και μετά μπήκατε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες του κανονισμού που δεν λειτουργεί, αλλά τελικά μας περιγράψατε την τραγωδία της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα αποθέματα. Αλλά κατά τη γνώμη σας, ε, τι θα πρέπει να γίνει. Σαφώς και δεν εκτιμάτε τον κανονισμό. Αλλά ποια είναι η λύση κατά τη γνώμη σας. Και τελευταία ερώτησή μου αφορά τα σχέδια διαχείρισης. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και τα 25 είναι σε επίπεδο κρατών μελών μόνο προβλέπονται σχέδια διαχείρισης ε, της Ένωσης ε, που θα έρθουν στο Κοινοβούλιο για συναπόφαση. Μάλιστα. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Έχει ερωτήσεις για όλους. Λάβετε φάγετε. Ποιος θέλει λοιπόν να απαντήσει. Μάλιστα, ο κύριος Τουδέλα πρώτα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να απαντήσω η κυρία Φράγα. Ότι ναι, δυστυχώς πιστεύουμε πως αυτές οι διατάξεις περί απορρίψεων στην Μεσόγειο, αυτός ο κανονισμός δεν είναι ο κατάλληλος και δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος και μόνο και μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους. Επειδή υπάρχει κίνδυνος να προωθηθεί η μαύρη αγορά σε νεαρά ψάρια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και αυτό το τονίσαμε όταν συζητιόταν ε, ο κανονισμός. Δυστυχώς λοιπόν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το μέτρο που υιοθετήθηκε. Και η δική μας δέσμευση είναι να βελτιώσουμε την επιλεκτική ανθεκτικότητα στην ε, Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πως είναι απαραίτητο. Πρέπει να μειωθεί η προσπάθεια και αυτό σημαίνει περισσότερη ε, δυνατότητα επιλογής, ε, διαχείριση και ανάκτηση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο. Δηλαδή απλώς κοινή λογική. Περί αυτού πρόκειται. Έχοντα όλα αυτά υπόψη, πιστεύουμε πως ορισμένα μέτρα έχουν υιοθετηθεί, όπως για παράδειγμα η απέτηση για εκφόρτωση των νερών ψαριών σε είδη, είτε είναι μήνυμο μεγεθών είτε όχι. Αυτό το μήνυμο μέγεθος θα αποτελέσει το μέγεθος αναφοράς στην εκφόρτωση και η εκφόρτωση θα είναι υποχρεωτική. Ένα τέτοιο μέτρο είναι απαραίτητο διότι πιστεύουμε πως χρειάζεται να εξετάσουμε ποιος μηχανισμός πρέπει να εισαχθεί ώστε να παρεμποδίζονται τέτοιου είδους εκφορτώσεις οι οποίες στην ουσία τροφοδοτούν την μαύρη αγορά και όπως και σε άλλες περιοχές στη Μεσόγειο τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικά πολύτιμα από οικονομικής άποψης. Ναι, πιστεύουμε ότι η συνδιαχείριση είναι κάτι το οποίο δεν είναι νέο. Όλοι γνωρίζουμε τη συνδιαχείριση, η οποία υπάρχει σε κάθε εγχειρίδιο διαχείρισης αλληλείας εδώ και 40 χρόνια. Αλλά ίσως ο τρόπος εφαρμογής του με κάποιον καινοτόμο τρόπο είναι που λείπει. Να το βάλουμε δηλαδή σε, κάποιο, ε, σε κάποια βάση ε, και να επεκταθεί η Επιτροπή των ε, φορέων και σε επιστήμονες. Δηλαδή είναι ένας τρόπος αυτός για να προχωρήσουμε. Ένας από τους τρόπους. Θα είμαστε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί βέβαια. Γιατί δεν υπάρχει μια συνταγή για να βγούμε από μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Καταστροφική θα έλεγα. Πάντως εμείς αυτό προτείνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε ε, δει ότι τα αποτελέσματα εκεί που έχει δοκιμαστεί η διαχείριση είναι πολύ θετικά. Έχουμε την ε, Λία Σεντίδο στην Ισπανία, στην Καταλωνία και έχουμε και άλλη μια εμπειρία που είναι μια υπόθεση όπου υπάρχουν και τράτες για τα βαθυπελαγικά ήδη. Δηλαδή η συνδιαχείριση δεν αφορά μόνο την μικρή κλίμακα αλληλεία, αλλά μπορεί να ε, ταιριάζει και για άλλου είδους ε, αλληλεία, γιατί επιτρέπει τον συνδυασμό των αναγκών σε συγκεκριμένα τοπικά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα ε, χειραφετεί τους αλληλείς, τους επιτρέπει να αισθάνονται ότι είναι μέρος της λύσης, ότι μπορούν να αναλάβουν τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται, γιατί τα έχουν συν στην ουσία, απλοποιούνται οι έλεγχοι και αυτό αυξάνει και τη συμμόρφωση. Οπότε τουλάχιστον αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκαγιάρ ή Μπομφίλιο. Nosotros, claro, órgano de cogestión, Μάλιστα διαχείριση ή σώματα διαχείριση, όπως και αν το πούμε, πιστεύουμε πως τέτοια σώματα έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν, είναι σημαντικό να τους ακούσουμε κιόλα. Δεν έχει σημασία πώς θα το αποκαλέσουμε. Εγώ στηρίζω την χρήση τέτοιων σωμάτων. Ο κύριος Μπονφίλιο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και Όσον αφορά την Ιταλική ελία και την ε, Διαχειριστική Επιτροπή, μια διαχειριστική επιτροπή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα πιστεύω πως είναι ένας από τους δρόμους της διεξόδου που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γιατί ίσως να είναι και αυτός ο τρόπος που ε, μάλλον στη Μεσόγειο μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό γιατί όταν πριν έλεγα ότι κάτι δεν πάει καλά αυτό προκύπτει από ένα κεντρικό στοιχείο το οποίο μας ε, παρουσίασε και ο δόκτωρ Όσιο σήμερα, αλλά ίσως μην το παρατηρήσαμε αρκετά. Είμαστε πρώτη φορά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας, αλλά αυτό δεν προκαλεί μείωση της θνησιμότητας των αλλιευμάτων. Βεβαίως, το μείγμα των τεχνικών μέτρων από τον οποίο αποφασίστηκε η παρέμβαση μέχρι τώρα δεν αρκεί. Ίσως να χρειάζεται να πούμε, ίσως μάλλον πολύ νωρίς να πούμε ότι δεν λειτουργούν αυτά τα σχέδια τα διαχειριστικά. Ίσως πάντως ούτε τα τεχνικά μέτρα είναι ίδια για όλους, μπορούν μάλλον να είναι ίδια για όλους ούτε τα διαχειριστικά σχέδια να χώρα για ένα σύστημα ληφτικό πρέπει να βρεθούν μορφές διαχείρισης που να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και μέσω από μικτές διαχειριστικές επιτροπές όπως έλεγε πριν ο, φίλο, φίλος ε, του Ντέλα. Νομίζω πως αυτό είναι ο σωστός δρόμος αλλά και άλλα πολλά πρέπει να γίνουν η επιλεκτικότητα είναι μια πτυχή, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πως ε, είναι και αυτό έχει περιορισμούς τεχνικού τύπου. Ε, αλλά όλα αυτά δεν ωφελούν αν πάμε στην Μεσόγειο να ψαρεύουμε νερό γιατί δεν υπάρχουν μεγέθη τα οποία να δικαιολογούν την οικονομία ενός αλλιευτικού σκάφους 250 ε, ε, τόνων που βγαίνει στη θάλασσα, γιατί θα είχε αρνητικό, θα έχει ζημιά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε σε τοπικό επίπεδο, σε κάθε GSA, δηλαδή ένα συνδυασμός ανάμεσα στο σχέδιο ανά ανα-GSA και σχέδιο ανά σύστημα ε, θα μπορούσε να είναι ένας δρόμος. Πολλά μπορούν να γίνουν και στη γη. Ε, πολλά, πάντα σκεφτόμαστε τη θάλασσα, αλλά εγώ θυμάμαι πάντα ότι ο Αλιάς δεν ψαρεύει τίποτα το οποίο να μην αποφέρει κάποιο αντίτιμο στην αγορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους καταναλωτές και με την αγορά πριν να πούμε για το τι θα γίνει στη θάλασσα. Γιατί είναι προφανές ότι αν ένα είδος δεν το αγοραζόταν θα είχαν το ενδιαφέρον του. Και εδώ δεν δουλεύουμε αρκετά. Βέβαια, πρέπει να προχωρήσουμε με μια ολόκληρη μορφή, μάλλον για την αντιμετώπιση της παράνομης αλληλείας. Γιατί υπάρχει, δεν μπορούμε αυτό να το αρνηθούμε. Θα πρέπει να υπάρξει διάκριση για την παράνομη αλληλεία, την επεισοδιακή, σποραδική, εποχιακή που δίνει τη δυνατότητα για να καλύψει κανείς κάποιες τρύπες από την πειρατική παράνομη αλληλεία που γίνεται επιμονή μου βάσεως. Πρέπει λοιπόν να γίνει διάκριση ανάμεσα στις διάφορες αυτές μορφές παράνομης αλληλείας. Θα πρέπει να δούμε την περιφερειοποίηση που μας δίνει μια άλλη ευκαιρία και Πιθανώς μέσα στην αναζήτηση ενός νέου τρόπου που συνδυάζει διάφορες τεχνικές διαχείριση θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Πέρα δηλαδή από την επιλεκτικότητα, εγώ ανησυχώ πάντοτε για την, ε, την ε, επιβίωση του στόκ ανανέωσης, δηλαδή των γεννητόρων ε, πρέπει να προστατεύσουμε και τα μεγάλα μεγέθη, όχι μόνο τα μικρά, με συγκεκριμένη στοχευμένη πολιτική και ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ζώνες αναπαραγωγής και εκεί δεν βρίσκονται πάντοτε οι, ε, τα ψάρια που είναι σε ηλικία αναπαραγωγής, πάνε μόνο σε συγκεκριμένες εποχές. Σε μια θάλασσα λοιπόν όπως η Μεσαίγειο μπορεί κανείς να τη θεωρεί μια μικρή λίμνη, αλλά είναι περίπλοκη αυτή η λίμνη είναι μια λίμνη που πρέπει να παρέμβουμε και με το... Ε, και με το τον ε, με τον ιστέρι πολύ προσεκτικά δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ρίχνουμε τσεκουριές ε, με το μπέλεκι. Ε, σας ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα κάπως. Άλλος που θέλει να λάβει το λόγο, αν δεν υπάρχει ένας άλλος. Νομίζω ότι... Α, εκεί, παρακαλώ. Κομισιόν. Πρόεδρε, η ερώτηση κυρία Λέβιν για τα σχέδια διαχείριση. Υπάρχει δυνατότητα για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράση. Προβλέπεται στον κανονισμό. Όμω, προ το παρόν, προκρίναμε μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω, γιατί αυτή είναι και η φιλοσοφία του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Όπως γνωρίζετε, στη Μεσόγειο υπάρχουν περιορισμένες αποκλειστικές ζώνες. Πρόκειται για χωρικά ύδατα δηλαδή. Άρα ξεκινάμε από τα κρατημέλη, τα οποία ορίζουν τα εθνικά σχέδια δράσης και το λεφτό προς απάντηση και του προηγούμενου σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές δημορφίες. Αυτή είναι η προσέγγιση. θέλαμε τώρα να συνδέσουμε αυτήν την προσέγγιση πρώτον με την αποτελεσματικότητα των σχεδίων και δεύτερον με την διαδικασία περιφερειοποίησης όπου τα κρατημέλη μαζί με το Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα το ΡΑΚ να υποβάλουν σχέδια σε υποπεριφερειακό επίπεδο. Ας πούμε για την Αδριατική ή έστω για την Βόρειο Αδριατική ή για τον κόλπο του Λέοντα κλπ. κλπ. Για συγκεκριμένες περιοχές όπου τα αποθέματα ουσιαστικά τα μοιράζονται κάποιες χώρες όπου χρησιμοποιούνται λίγο πολύ τα ίδια αλληλευτικά εργαλεία. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες εκπόνησης διασυνοριακών σχεδίων στο πλαίσιο της νέας αλληλευτική πολιτική όσο και στο πλαίσιο του κανονισμού. Η δυνατότητα λοιπόν υπάρχει. Παραμένει ανοιχτή και είναι και κάτι το οποίο θα προωθήσουμε τους επόμενου μήνε στο πλαίσιο και στην πορεία της λεγόμενης περιφερειοποίησης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή την ακρόαση. Νομίζω πως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική και ευχαριστώ και πάλι όλους όσους ε, όλους τους εισηγητές. Ωστόσο, μένουν διάφορα, μας δίνει μάλλον τροφή για σκέψη αλλά και χώρο για συμβιβαστικές λύσεις που θα πρέπει να, να υιοθετήσουμε και σκέφτομαι την Κομισιόν, αλλά βεβαίως τονίστηκε και, και κάποιες συνέπειες που ήδη είχαν ε, πει κάποιοι, είχαν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απορρίψεις και τα προβλήματα που θα μπορούσαν εδώ να προκύψουν, όπως φάνηκε. Κλείνω πάντως λέγοντας ε, το εξής που είπε ο κύριος Μπονφίλιο ότι δηλαδή η μεταρρύθμιση θα μας ε, προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία και θα πρέπει αυτήν να την εκμεταλλευτούμε ώστε να κάνουμε πραγματικά και στην Μεσόγειο ε, να λάβουμε τέτοια μέτρα ώστε η αλληλεία να είναι βιώσιμη. Και όταν λέω βιώσιμη, όχι μόνο να υπάρχουν ε, ε, τα είδη, αλλά να επιβιώσουν και οι ελευτικοί μας κλάδοι με τόσο κόσμο που εργάζεται εκεί. Σας θυμίζω τις 6.30 είστε προσκεκλημένοι. Νομίζω πως έχουμε ισπανικά προϊόντα στη δεξίωση που είναι πάντοτε καλά στον πέμπτο όροφο του κυρίου Σκτηρίου. Αύριο συναντήσουμε στις 9 με τους συντονιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστεί και τους διερμηνείς ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εμείς και μας προσκαλεί και στο, στη δεξίωση.